Αν έχετε την καλοσύνη να καθίσετε, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας λοιπόν. Σας καλωσορίζουμε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ε, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε κατά τα επόμενα πέντε έτη. Ε, για την Επιτροπή αυτή που είναι μια μικρή επιτροπή αλλά έχει πάρα πολλά θέματα που ε, είναι στην αρμοδιότητά της κλιματική αλλαγή, δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μονίμως κατά νου ότι οι δράσεις που αποφασίζουμε εδώ επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων και να έχουμε τη μακριά προοπτική κατά νου ε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προστατεύσουμε τα αλληλευτικά αποθέματα αν θέλουμε να έχει μέλλον η αλληλευτική βιομηχανία αλλά πρέπει να έχουμε και τη μεγάλη εικόνα και τη μικρή, τα πιο μικρά, τα καθημερινά έτσι ώστε να ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις πρώτες ύλε, τα ψάρια σε αυτό το τομέα, αν θέλουμε να ευημερήσει. Λοιπόν, πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, προτείνω να εγκριθεί. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Το δεύτερο θέμα, πρέπει να σας πω, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και αφορά τον κύριο Μπράτφορντ, ένα νέο συνάδελφο από την Πορτογαλία, από τις Αζόρες συγκεκριμένα, που θα ερχόταν κοντά μας, αλλά μας ενημέρωσαν για την αποβίωσή του την προηγούμενη εβδομάδα ε, και πρέπει να, πάω, πρέπει να πω ότι χαιρόμουν πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συνέβη και με την έγκρισή σας εκ μέρους της Επιτροπής θα στείλω μία συλληπιτήρια επιστολή στην οικογένειά του propose now the adoption of the minutes of the constituent constitutive how do you pronounce that the set up meeting <laughs> of the 10th of July. Λοιπόν, ε, συστατική η Επιτροπή έγινε στις 10 Ιουλίου, Ε, εγκρίνονται τα πρακτικά της Επιτροπής αυτής και τώρα περνάμε στο σχέδιο προϋπολογισμού Όταν ανέλαβα την Προεδρία, η Γραμματεία μου παρουσίασε το σχέδιο προπολογισμού. Και λίγο πολύ, αυτό είναι και το έγγραφο που κατατέθηκε και σε εσά, είναι μία γνωμοδότηση που υποβάλλουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και ε, βεβαίως η γνωμοδότηση αυτή είναι ανοιχτή για τις προτάσεις σας ε, μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι. Δεν ξέρω πού είναι ο εκπρόσωπος. Α, είναι εκείνη η εκπρόσωπος της ε, Κομισιόν. Η κυρία Ντόρι Καρέιρα. Κυρία Καρέιρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή και πάντα χαρά για μένα το ότι βρίσκομαι και πάλι σε αυτή την Επιτροπή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχόμενοι σε όλους σας τα καλύτερα για αυτή τη θητεία. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα επίμαχο θέμα που είναι το σχέδιο προεπλογισμού για τον 2020. Γιατί το 2020 είναι η τελευταία χρονιά αυτή τη οικονομική περίοδου, γιατί όπω όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, συζητάμε ήδη τώρα ε, τον προεπλογισμό για την ε, περίοδο 2021. 21-27. Άρα δηλαδή η επόμενη χρονιά είναι μια χρονιά που είναι σημαντική για να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε αυτά που έχουμε επιτύχει και να εκπέμψουμε ένα ηχηρό μήνυμα όσον αφορά την εφαρμογή. Την εφαρμογή κατά την αμέσως επόμενη οικονομική περίοδο. Όσον αφορά λοιπόν ε, στα θέματα αλίας, και θαλάσσιων θεμάτων. Προτείνουμε κάποια ποσά. Όσον αφορά τις ε, πιστώσεις υποχρεώσεων, αυτά που έχουμε δεσμευτεί για το 20 και τα επόμενα ετή, η Κομισιόν προτείνει πάνω από ένα δις ευρώ. Και όσον αφορά τις ε, πιστώσεις πληρωμών, για να μπορέσουμε να ε, τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας από πέρυσι, προτείνουμε 960 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα κονδύλια καλύπτουν τρία πράγματα. Καλύπτουν τα ταμεία, τα ευρωπαϊκά ταμεία αλίας και θάλασσας καλύπτονται οι διεθνείς οργανισμοί αλίας και θάλασσας και επίσης και οι φορείς ελέγχου στο Βίγκο. Και κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για κάθε ένα από αυτά τα τρία διαφορετικά στοιχεία. Βεβαίω, οι περισσότερε δαπάνε είναι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα και Αλία, η MFF. 90% είναι με κοινή διαχείριση που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία ε, φροντίζουν για την ε, χρήση αυτών των κονδυλίων. Έτσι λοιπόν για τα επόμενα έτη προβλέπουμε τη συνεχιζόμενη εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων και προτείνουμε 858 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά βέβαια εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχουμε πάρα πολύ αυστηρά στην Επιτροπή. Και εδώ έχω ευχάριστα νέα για εσά. Όπω ξέρετε, το ταμείο αυτό, το EMFF, ξεκίνησε πολύ αργά το 2014, αλλά τώρα όμω με βάση την έκθεση εφαρμογή του προηγούμενου χρόνου, ε, στα κράτη-μέλη επιταχύνεται η διαδικασία 33.000 προγράμματα έτρεχαν πέρυσι στα κράτη-μέλη, δηλαδή διπλάσιος αριθμός ε, σε σχέση, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, το 2017. Ε, η συνολική αξία αυτών των προγραμμάτων είναι 5 δις ευρώ και το ίμιση καταβάλλεται από αυτό το ταμείο, που σημαίνει ότι περίπου το ίμιση του EMFF, ε, των κονδυλίων για τον EMFF, ε, πλέον έχουν δεσμευτεί και επίσης και εκταμιευτεί. Αυτά όσον αφορά τη διαχείριση. Ε, το 90% του Ταμείου από τα κράτη-μέλη, το 10% το διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως για θαλάσσια πολιτική και συνοδευτικά μέτρα για την εφαρμογή της αλληλευτικής πολιτικής, όπως είναι οι ε, επιστημονικές συμβουλές. Για το 2020 έχουμε βασιστεί στον προγραμματισμό καταρχήν εντοπίζοντας τις ανάγκες και σεβόμενοι πλήρως ε, την ε, θεματική κατανομή στο Ταμείο αυτό με βάση τον κανονισμό. Πάμε στο δεύτερο ήμιση του προϋπολισμού, εκεί όπου πρόκειται για την στήριξη των συμφωνιών και των περιφερειακών αλληλευτικών οργανισμών. 142 εκατομμύρια ευρώ ζητάμε για την επόμενη χρονιά. Το ποσό αυτό καλύπτει βέβαια τις συμφωνίες αλίες που ήδη εφαρμόζονται, αλλά και εκείνες οι οποίες προβλέπεται ότι θα εφαρμοστούν το 2020, όπως παραδείγματος χάνε αυτή με το Μαρόκο, γιατί μόλις τώρα προέκυψε η επικύρωση από τις αρχές του Μαρόκου. Επίσης, ε, προβλέπουμε να καλύψουμε ε, τις συμφωνίες που ανανεώθηκαν το 2019, όπως είναι αυτή με την Γουνέα Μπισάου ή το 2020 σε Ιχέλε, παραδείγματο χάρη. Ενδεικτικά τα λέω. Άρα δηλαδή σε αυτό το τμήμα του προλογισμού δεν έχουμε πολλά χρήματα για να δαπανίσουμε και έχουμε όμως κάποια χρήματα, ένα απόθεμα στον προπολογισμό για τις επιτυχίες που έχουν, για τις συμφωνίες μάλλον που έχουν κριθεί επιτυχημένες. Τον φορέα στο Βίγκο, τον ε, Ευρωπαϊκό Φορέα Ελέγχου έχουμε προτείνει 16,7 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο συμβαδίζει με τη συμφωνία που έγινε ε, ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τον κανονισμό ακτοφυλακής ΕΦΚΑ και ΕΜΣΑ. Αυτός είναι ο κανονισμός, η συμφωνία που έχει επιτευχθεί. Και αυτά προστίθενται στη βασική δουλειά του φορέα που είναι ο έλεγχος και η εφαρμογή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Όσον αφορά τώρα τις ε, προκατακτικές δράσεις και τις διμερείς συμφωνίες, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αυτή μας κατέθεσε μια πρόταση για πιλωτικά προγράμματα. Το εξετάζουμε και θα επανέλθουμε επ' αυτού σύντομα. Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζουμε με τη γνωμοδότηση, απλά να έχετε κατά νου ότι όσον αφορά το δικό μας τον προϋπολογισμό για την Ελία, ε, κατά 4 εκατομμύρια κόπηκε ο προπολογισμό ε, από το Συμβούλιο και γι' αυτό ε, θα χαιρόμασταν αν το Κοινοβούλιο μας στήριζε στη δική μας την αρχική πρόταση. Πολύ ευχαρίστω να σας απαντήσω αν έχετε να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε πρώτα τους ε, συντονιστές, ο κύριος sombrero. Κοιτάξτε, έχω διπλή ιδιότητα συντονιστής, αλλά και αντικαθιστώ και την κυρία εισηγήτρια, η οποία δεν μπόρεσε να προσελθεί για προσωπικούς λόγους. Έχω εδώ την παρέμβασή της, μου ζητούσε. Εγώ μπορώ να παρέμβω πρώτα αν επιτρέπεται ως σκιώδης λοιπόν αντικαθιστώντα της και μετά ως συντονιστής. Θα κάνω και τα δύο. Η κυρία Μοντέιρο de λέει το εξή. Είναι η σκιώδης εξ ονόματος ομάδας μας. Η πρόταση για τον προϋπολογισμό της φαίνεται ισορροπημένη, ότι καλύπτει τα πιο σημαντικά, τα υδατοκαλλιέργεια, ε, μικρή κλίμακα το θέμα του Βίγκο και το θέμα του Brexit ευθυγραμμίζεται μετά του Πρόεδρου Ντέιβις και ότι η πολιτική αλληλείας μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μόνο με επαρκή στόχους ε, που θα προστατεύουν και την απασχόληση χιλιάδων ανθρώπων. Πρέπει να πολεμήσουμε για μια πληρέστερη επιστημονική γνώση και κάλυψη για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καλύτερα. Επίσης θα πρέπει να ε, τονίζεται ε, μια επαυξημένη προστέμενη αξία για τις ε, παράκτιες ζώνες μας και δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ τους άνδρες και τις γυναίκες που ζουν από τη θάλασσα και την οικονομία της. Τώρα για μικρές τροποποιήσεις οι προϋπολογισμοί πρέπει να ευθυγραμμίζεται προς τους στόχους αυτούς και λέει η κυρία Γιλιάρ να προσφέρουν ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών στόχων της πολιτικής αλίας. Το σύντομο κείμενο που μου έδωσε η κυρία Γιλιάρ είναι αυτό. Ε, ο εγώ ο ίδιος, να πω ότι συμφωνώ με την πρότασή της, Πρόεδρε, και θα υπέβαλα δύο σύντομες τροπολογίες. Πρώτον, για να τονίσουμε την σημασία με, τους, ε, με τις βιώσιμες συμφωνίες με τρίτες χώρες για την αλία, που επιφέρουν και μια πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Σήμερα επιστρέφουμε στο Μαρόκο ως ευρωπαϊκό στόλος και αυτό είναι ένα από, τις, ένα από τα καλά σημάδια της συμφωνίας αυτής και να επιμείνουμε επίσης εν ώψη του προϋπολογισμού για την περιοδο 2021 2021-2027 πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους για την αλία, αυτό έχουμε ανάγκη και για την ε, περίπτωση του Brexit αυτό δεν πρέπει να είναι εμπόδιο ώστε ο προϋπολογισμός μας να εξακολουθεί να είναι φιλόδοξος. Ευχαριστώ. Τι εννοείται όμω με την ανηφιλόδοξου εδώ. Εκτό μικροφώνου. Α, ε, να μην έχουμε περικοπές. Όπως είναι η πρόταση που έχουμε στο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Αλλά να ενισχύουμε αυτήν την ε, οικονομική διάσταση. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο σκιώδης της ομάδας μας είναι ο κύριος Κόρμπετ. Ήθελα απλώς σύντομα, ε, συμφωνώ με τον πρόεδρο για τον προϋπολογισμό, ήθελα απλώς να υποβάλω μια ερώτηση στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, της Κομισιόν. Είχαμε ένα πρόβλημα εκτέλεσης του MFF για τα εθνικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία ενεκρίθησαν ε, καστηριμένα και η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών των επιχειρησιακών ήταν αργή. Μας λέει εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι αυτά κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, καλώς. Ε, μας λείπει ένας χρόνος, ενάμιση για να ολοκληρώσουμε το πλαίσιο αυτό, αλλά μας έδωσε κάποια στοιχεία, αλλά θα ήθελα να καταλάβω ποιο είναι ακριβώς το ποσοστό εκτέλεσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων μέχρι στιγμής. Ανέφερε κάποια μεγέθη ότι είμαστε περίπου στο 50%, δεν ξέρω αν έτσι ακριβώς είπε, αλλά θα ήθελα πιο λεπτομερώς να καταλάβω την ποσόστοση δαπανών, δηλαδή εκτέλεσης των εθνικών επιχειρησιακών Επίσης αναφέρθηκε η εκπρόσωπος της Κομισιόν σε μια περικοπή 4 εκατομμυρίων και εμεί ζητούμε ο πλευράς Κοινοβουλίου είναι να επανέλθουν οι πόροι αυτοί. Πάντοτε στο Κοινοβούλιο ε, όταν υπήρξαν περικοπές ζητούσαμε να επιστρεφούν οι πορεία, αλλά θα ήθελα να μας πει η, η εκπρόσωπος της Κομισιόν αυτή η περικοπή των 4 εκατομμυρίων εγώ δεν την είχα δει. Σε ποιο κονδύλι εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Αρκετά λεπτομερείς οι ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίω. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του EMFF, τα στοιχεία που σας ανέφερα στην αρχή ήταν το εξής. Το 45% του ταμείου έχει ήδη δεσμευθεί προς εκταμείευση συνολικά. Τώρα, για τις ε, πληρωμές που έχουν γίνει όντως, βρισκόμαστε στο 23%. των πόρων που έχουν δαπανηθεί. Ε, για να συγκρίνουμε με άλλα ταμεία, το Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη. βρίσκεται στο 28%. Το Κοινωνικό Ταμείο βρίσκεται στο 30%. Θεωρούμε ότι είναι αρκετά καλά λοιπόν τα στοιχεία, γιατί όπως ξέρετε ξεκινήσαμε ένα χρόνο αργότερα περιμένοντας ε, την ε, υιοθέτηση της νομικής βάσης. Και όπως ε, είπατε, και τα επιχειρησιακά προγράμματα άργησαν να υλοποιηθούν από τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν είναι τα συνολικά στοιχεία για τα 27 κράτη-μέλη, πλην του Λουξεμβούργου που δεν διαθέτει τέτοιο πρόγραμμα. Και βέβαια υπάρχουν και διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Όμως σας λέω συνολικά ποια είναι τα στοιχεία. Και όταν είπα ότι έχουμε ήδη επιταχύνει το λέω επειδή μέσα σε ένα χρόνο έχει διπλασιαστεί η εκτέλεση του προπολογισμού. Α, για τα 4 εκατομμύρια. Υπήρξε αυτή η περικοπή στο SFPA, δηλαδή στο τμήμα του προπολογισμού που αφορά τις ε, συμφωνίες τερικής σχέσης ε, και στην γραμμή για τα αποθέματα. Τα κονδύλια λοιπόν που έχουμε αφήσει κατά μέρο για συμφωνίες τις οποίες διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή και περιμένουμε να δεχθούν σε ισχύ του χρόνου και ίσως το Συμβούλιο είναι λίγο λιγότερο αισιόδοξο από ότι εμείς. Θεωρούσαν λοιπόν ότι μπορούν να βγάλουν αυτά τα 4 εκατομμύρια. Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να τα δαπανίσουμε και γι' αυτό θα θέλαμε να επανέλθει αυτό το κονδύλι στο αποθεματικό. Κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για το 29% για την τεχνολογία και τον εξοπλισμό μας προβληματίζει λίγο. Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για την εκφόρτωση και χαμηλότερε υποχρεώσει. Και μια επιστημονική προσέγγιση είναι σημαντική σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και υλοποίηση πολυετών ε, σχεδίων. Ε, φυσικά έχουμε και τροπολογίες προς αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Κόντε. Κολέα Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά ε, τις ε, δαπάνες για τη θέματα έρευνας, νομίζω ότι τα κονδύλια θα πρέπει να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο. Εμείς ε, θα υποβάλουμε προτάσεις που θα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικο-οικονομικό στοιχείο και αναφέρομαι κυρίως στο πόσο σημαντική είναι η μικρή στόλη. Είναι περίπου το 50% των σκαφών, ληφτικών σκαφών που έχουν καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου το ίμιση δηλαδή. Θα πρέπει Πρέπει λοιπόν ε, και σε αυτή την ε, αλία και στη μεταπητική, τη μικρή αλία, να διατεθούν ε, περισσότερα κονδύλια για να διευκολύνουν την εκφόρτωση και για να προάγουν και την διαφοροποίηση της οικονομίας, να προάγεται η αλία και ο τουρισμός. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής οικονομική ενίσχυση, να υπάρχουν ικανοποιητικά κονδύλια, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας περιορισμός στη δραστηριότητα των αλίων. Και θα ήθελα να πω ότι οι αλλοίς ε, δεν είναι μόνο εκείνοι που ενδιαφέρονται για τα αποθέματα και αυτοί θέλουν προφανώς να διατηρήσουν την πρώτη ύλη. Έχουμε την διαφοροποίηση στη βιομάζα, στην κλιματική αλλαγή, έχουμε την ε, ρήπανση. Αυτά είναι, ένα από τα μεγαλύτερα, είναι μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν, όπως σας είπα, να υπάρχει και κάποια, σε σε κάποια εναρμόνιση ε, το Ισαλίας με το περιβάλλον. Ε, έχουμε κατά νου τις πλαστικές ε, ύλες που υπάρχουν στη θάλασσα. Μην ξεχνάμε το πόσο σημαντική είναι η θάλασσα για τους αλείς μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή κονδύλια που να εκταμιεύονται και για συμβουλευτικές ε, δραστηριότητες οι συμβουλευτικές αυτές δραστηριότητες ε, είναι από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την περιοχή και διαδραματίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές ε, που χαράσσονται και που υπάρχουν στα δικά μας τα πολιτή προγράμματα. Θέλω επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει όσο μεγαλύτερη απλούστευση του ΦΕΑΠ έτσι ώστε να είναι δυνατόν να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση να βελτιωθεί η κατάσταση των αλλίων ε, και Τέλος, ε, μην ξεχνάμε ότι το Brexit ε, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις ε, στην Αλία, κυρίως στο ΦΕΑΠ. Αν λοιπόν δεν υπάρχουν οικονομικές, ικανοποιητικές προβλέψεις, νομίζω ότι υπάρχουν και απόλυτες συνέπειες. Thank you for your comments. Uh, Mrs. Dodds. Κυρία Dodds. Thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά το IMFF, e είπατε ότι ε, το 40% των κονδυλίων έχει δεσμευτεί, το 23% έχει εκταμιευθεί. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα πώς ε, δαπανώνται αυτά τα κονδύλια ε, σε ό,τι αφορά την στήριξη των παράκτιων κοινοτήτων σε σχέση με τη βιώσιμη αλληλεία και τα επιστημονικά προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να κινηθούμε προς ε, μια πιο βιώσιμη αλία στο μέλλον. Αναμενόμενο είναι το ότι θα αναφερθώ στο Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο αύριο, από αύριο και μετά θα έχει νέο Πρωθυπουργό. Όποιος και αν είναι αυτός, έχει αναφέρει ότι θα φύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου. Άκουσα μεγάλη προσοχή τα όσα είπατε για το έτθα και δεν βλέπω πώς ακριβώς προτίθεστε να στηρίξετε την αλληλεία σε περίπτωση μη συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να τηρεί μία σκληρή στάση και από την άλλη έχουμε και μια κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο που θεωρεί απαράδεκτο το backstop, υπάρχει πραγματικά πιθανότητα να φύγει χωρίς συμφωνία το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμώ, το έχω πει πολλές φορές, ότι πρέπει να φύγουμε με συμφωνία και όλα να είναι καλά οργανωμένα. Όμως με ενδιαφέρει να δω πώ ακριβώς ε, θα εξετάσετε το ΕΤΘΑ, πώς υποστηρίξετε την αλία. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανακτήσει έλεγχο των θαλασσών του και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν διαπραγματεύσει και συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό θα έχει επιπτώσεις ενδεχομένω και για την ε, Ευρωπαϊκή Αλία. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι έχει σημειώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ερώτημα. Θα ακούσουμε μερικέ ερωτήσει ακόμα πριν τις απαντήσει. Η κυρία Σάιπίρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με το τελευταίο ερώτημα για τον Brexit και εσεί από την Αγγλία κατάγεστε. Αλλά και για τη χώρα μου, την Ολλανδία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και έχουμε στείλει και ω ΕΛΚ μια επιστολή για αυτό το θέμα. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με το ερώτημα. Μετά, το 45% και το 23%. Τι ακριβώς είναι αυτά τα ποσοστά που αναφέρατε. Και κάτι άλλο που, για το οποίο θα καταθέσω και τροπολογία, δεν πρέπει τώρα να κάνουμε έρευνα για την έρευνα. Είναι πράγματα που ήδη υπάρχουν. Το θέμα είναι ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε. Η μεγάλη, η μικρή, η στο κλίμα και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή οι αλληλείς στις 100 ε, χώρες έχουν ε, τα αριθμητικά στοιχεία. Αλλά μετά τα μεγάλα πανεπιστημία θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν έρευνα και άλλη έρευνα, ενώ οι αλληλείς ήδη έχουν τα στοιχεία έτοιμα. Και θα πρέπει και εμείς να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ευχαριστώ. Mr. Ferreira. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα όσα μας είπε. Θα ήθελα να πω σε ό,τι αναφέρθηκε για τον προπολογισμό, ε, διαφωνώ με τα όσα ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς δεν συμφωνούμε ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ικανοποιητική την κατάσταση σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ε, πιστώσεων ε, και εκταμιεύσεων. Όλα οι παράγοντες που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως είναι σημαντικοί και τους ε, συνεκτιμούμε. Όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και όλα αυτά βασίζονται στο γεγονός ότι το Ταμείο έχει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Πρέπει να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα όμως που αντιμετωπίζει και ο ίδιος ο Αλιέας. Καθώς λοιπόν προχωρούμε προς το τέλος ε, της πραγματικής περίοδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντί να προσπαθεί να, να οροποιήσει την κατάσταση και να μας ε, καθησυχάζει, να μας πει ότι όλα βαίνουν καλώς, Ίσως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να αφαιρεί κάποια προγράμματα από την τρέχουσα και να τα προσθέτει στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Γιατί δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους και δεν έχουμε προβλέψει και πολλά για την επόμενη περίοδο. Είδαμε λοιπόν τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο τέλος της προηγούμενη θητεία για το Ταμείο και καλό θα ήταν οι παρατηρήσει αυτές του Κοινοβουλίου να ληφθούν πλήρως υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά δεν χρειάζεται να απορρίπτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθεία ε, διάφορε προτάσει που έχει καταθέσει το Κοινοβούλιο. Μετά δεν ξέρω αν το έχει εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά είναι δεδομένο ότι δεν μπορούμε να εκδηλώσουμε την ικανοποίησή μας σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις μας προ το παρόν. Χρήσιμο λοιπόν θα ήταν σε αυτό το στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να σκέφτεται για την επόμενη πραγματική περίοδο, όπω είπα, και παράλληλα να προσπαθήσει να σκεφτεί και τι είδους προπαρασκευαστικές εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν. Μπορεί η Επιτροπή να προτείνει πιλωτικά προγράμματα, προπαρασκευαστικές ενέργειες. Είναι μια πρόκληση σε αυτό που μπορώ να απευθύνω προς την Επιτροπή. νέες ε, πιλωτικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες στις οποίες θα μπορούσε να προβεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρότι ξέρω δεν είναι η συνήθιση διαδικασία. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι γνώμη έχει για τα πιλωτικά προγράμματα που ήδη έχουν υλοποιηθεί σε αυτό το τομέα. Ένα μπορώ να σκεφτώ, ε, μέτρα στήριξης για την ε, μικρή κλίμακα και παράκτη αλία. Και εκεί, λοιπόν, υπήρξε ένα πιλωτικό σχέδιο. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας ε, ενημερώσει για το πώς προχωράει αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Και ολοκληρώνω. Αυτά θα ήθελα να ακούσω τι έχει να πει η Επιτροπή. Έχω ακόμα δύο για να κλείσω τον κατάλογο, έτσι. κυρία Ταντήρα, Ευχαριστώ πρόεδρε. Προφανώς ε, τα επαρκή χρηματοδοτικά μέτρα ε, στο τομέα της αλληλείας είναι ουσιώδες ώστε να επιτύχουμε τους στόχους της κοινή πολιτικής. Συμφωνώ με τις ε, κατευθυντήριες γραμμές γενικώ της πρότασης του Προέδρου. Θα προτείναμε κάποιες τροποποιήσεις ε, προς την κατεύθυνση και της ε, κυρίας Κόντε της εισηγητριάς μας αλλά θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία για κάποιες τροπολογίες που έχω την ε, πρόθεση να υποβάλω για τις παράκτιες ζώνες. Εγώ εκπροσωπώ την Σικελία και την Σαρδινία εδώ. Και υπό το φως προσφάτων διατάξεων που είναι ιδιαίτερα επιζήμιες για τις ζώνες αυτές, αναφέρομαι στον κανονισμό 982 τον σχετικό με τις διατάξεις για την αλληλεία στις περιοχές της συμφωνίας ε, CGPM που περιορίζει την αλληλευτική δραστηριότητα στις ζώνες Σικελίας αλλά και την WestMed που βελτιώθηκε σχετικά με την αρχική πρόταση της Κομισιόν αλλά προ... ενέχει ιδιαίτερα επιζημίες διατάξεις για την δική μας αλληλεία για τις δικές μας νήσους και επομένως ως προς τους στόχους βιωσιμότητας που είναι απολύτως σεβαστοί, ε, είναι πηγή οικονομικής ε, ανάπτυξης και απασχολησιμότητας ε, και πολύ σημαντικές για τα εδάφη και για τις περιφέρειες που ενέχονται. Ήθελα να υπογραμμίσω επίσης την κοινωνική διάσταση της πολιτικής αλίας για τις τοπικές κοινωνίες και για κάποιες παράκτιες και νησιωτικέ ζώνες που εξαρτώνται απολύτω από την αλληλευτική δραστηριότητα. Το εισόδημα πολλών νοικοκυριών εξαρτάται ακριβώς από αυτή την πηγή. Και πολύ συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα πρόσθετου κόστους ε, και μονίμων μείων εκτιμάτων που θα πρέπει να αντισταθμίζονται μέσω ε, των πρόσθετων πόρων του σχετικού ορισμού Ακόμα πιο σημαντικό εν ώψη προσφάτων διατάξεων που σα ανέφερα. Εμείς θα υποβάλουμε προτάσεις τροπολογίας υπό την έννοια αυτή και ελπίζω οι συνέλφοι να μπορέσουν να τι υποστηρίξουν. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Κύριος Μόντι, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Επιτροπής ε, για την ε, εισήγησή της. Εδώ έχουμε μία πρόταση ε, ψηφίσματος και στο κόμμα 3 ε, μιλούμε για τη διεθνή ύδατα και τις αποκλειστικές ε, ζώνες εκμετάλλευσης τρίτων χωρών. Εάν βέβαια συμβεί το Brexit, αυτή η ποσόστοση θα αυξηθεί. Και στο σημείο 3 και το 2 μιλούμε για επαρκείς ε, δημοσιονομικές προβλέψεις. Αλλά δεν ξέρω αν αναφερόμαστε και στο Brexit, συνυπολογίζουμε δηλαδή το Brexit και θα πρέπει να συστήσουμε ένα πι δελτα πι για την επόμενη περίοδο, αλλά δεν υπάρχει καμιά αναφορά, όπως είπε και η συνάδελφος, για το τι θα γίνει το 2020 και όχι στην επόμενη περίοδο. Και στην περίπτωση του Brexit μου κάνει εντύπωση που δεν υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Δηλαδή δεν έχουμε καμία πρόβλεψη προσαρμογής του προϋπολογισμού εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει. 31 Οκτωβρίου ή οποτεδήποτε ή και νωρίτερα δηλαδή. Και αν δεν έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη δεν θα ήταν φρόνιμο να προσθεθεί κάτι στην γνωμοδότηση αυτή ώστε να υπάρξει πρόβλεψη επαρκούς ε, ε, χρηματοδοτικής στήριξης για τις ε, αλίες εφόσον η Βρετανία αναλάβει την αλία. Μάλιστα θα ακούσουμε και την ε, πρόταση της Κομισιόν ο κύριος Ήτο. Ε, κοιτάξτε, εγώ θα κάνω μια παρέμβαση αν τους άλλους, δεν περιμένω να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν για να τοποθετηθώ. Εμείς, ε, εγώ εκπροσωπώ την Νουβέλα Κιτέν ε, και άλλες παρακτίες ζώνες και για τα κονδύλια που θα τοποθετηθούν στον προϋπολογισμό ε, πρέπει να έχουμε μια κινητοποίηση των περιφερειών αυτών ώστε ε, η χρηματοδότηση να είναι αποτελεσματική και λειτουργική όπως είναι σήμερα. Ε, εκμετα... με τη ευκαιρία για τη συζήτηση του προϋπολογισμού για τα υπέρ και τα κατά που αναφέρθηκαν να αναφέρω το εξής. Επί του MFF όχι για, ε, λάθος, για τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες διαπιστώνω ότι βεβαίως και πρέπει να έχουμε τέτοιες και βεβαίως και το πρόβλημα του Brexit αναπόφευκτα μας οδηγεί ακόμα περισσότερο σε αυτό, αλλά καλό θα ήταν ε, ε, να έχουμε γενικές ευρείες προσεγγίσεις. Δηλαδή εφόσον έχουμε έναν πόρο υδάτινο ο οποίος είναι κινούμενος και κινητός ε, και μιλώντας για τη Γουινέα Μπισάου ή την Μαυριτανία ακόμα και οι πόροι της ε, ε, άλλων περιοχών και άλλων χωρών μπορούν να επηρεάζονται από τις συμφωνίες αυτές και αν πράγματι υλοποιηθεί το Brexit ίσως θα, πρέπει να, ίσως θα χρειαστεί με τις χώρες αυτές ε, που απέρχονται να βρούμε μια κοινή συμφωνία για να διαχειριστούμε τους ελευθερικούς πόρους ε, με τρόπο υπεύθυνο. Είτε είναι μέλη δηλαδή της Ένωσης είτε όχι. Δηλαδή επανερχόμαστε σε μια ανάγκη ευρείας προσέγγισης. Και έχω και το εξή σχόλιο. Ε, μιλούμε για την Επιτροπή Αλίας εδώ. Αλλά μήπως είναι λίγο περιοριστικό αυτό. Γιατί ε, το πρόβλημα της αλίας είναι ε, ένα σημαντικό και ευρύτατο πρόβλημα. Μιλούμε για τους υδάτινους και αλλιευτικούς πόρους ε, και κακώς θα έπρεπε να εστιαζόμαστε μόνο στην αλληλευτική δραστηριότητα και το EMFF αφορά και στην υδατοκατελήρια και στη θάλασσα και στην αλία. Επομένως, ίσως αυτή η επιτροπή θα έπρεπε να λέγεται Επιτροπή Θαλασσών ή Οκεανών για να αναφερόμαστε στα οικοσυστήματα τα θαλάσσια, τα ωκεάνια, που είναι το πραγματικό πρόβλημα της ε, μείωσης των πόρων και της σωστής διαχείρισής τους. Πρέπει, ε, και πάλι επιμένω, πρέπει να είμαστε ευρύτεροι στην ε, προσέγγιση μας και να μην εστιαζόμαστε μόνο και μόνο σε μία αλλιευτική δραστηριότητα, η οποία όμως εξαρτάται από τους θαλάσσιους πόρους και τους ωκεάνιους πόρους. Thank you. I look forward to hearing your... Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις σε αυτήν την πρώτη ανταλλαγή. Επομένως, ρωτώ, ζητώ από την εκπρόσωπο της Κομισιόν να απαντήσει στα μέλη. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ πλούσια αυτή η συζήτηση και ξεκινάμε με το θέμα του Brexit, γιατί ετέθη από αρκετά μέλη. Ε, Βεβαίω ε, όλοι θεωρούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ε, θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση συντεταγμένα με βάση μια συμφωνία που θα έχει προηγηθεί. Αν δεν συμβεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και επίσης τον έκριναν και οι συνομοθέτες μία σειρά μέτρων ετοιμότητας που αφορούν και την αλία και τις ε, θαλάσσιες υποθέσεις. Εγκρίθηκαν αυτά στις 25 Μαρτίου. Ε, για μας αφορούν κυρίως δύο πράγματα. Από τη μια ε, προβλέπουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη που θα πληγούν περισσότερο, οι στόλοι που θα πληγούν περισσότερο από τη μη δυνατότητα πρόσβασης ε, σε ε, ύδατα της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου θα λαμβάνουν μία αποζημίωση οι αλής Αυτό είναι ένα από τα μέτρα τα οποία προβλέπουμε. Και ένα άλλο μέτρο είναι ότι θα αλλάξει το σύστημα αδειοδότησης να μπορούν δηλαδή οι να αποκτούν άδεια για να αλλιεύουν στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου ε, ως μιας ε, τρίτης χώρας. Αυτά τα μέτρα έχουμε αποφασίσει, υπάρχει πολλή ανασφάλεια, αλλά αυτά τα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, θα δώσουν κάποια ε, σιγουριά στους αλλοίς μας. Όσον αφορά τώρα άλλα θέματα που αφορούν στο ε, τι ακριβώς κάνει το Ταμείο, γιατί βεβαίως ε, σας ανέφερα αριθμούς, ε, αυτά είναι πολύ στεγνά, πρέπει να ξέρουμε τι επιτυγχάνει το Ταμείο. Βέβαια θα έπρεπε να μακρηγορήσω για να σας παρουσιάσω ένα λεπτομερή απολογισμό, αλλά αν συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε, να στείλω στη Γραμματεία μία έκθεση που καταρτίζουμε κάθε χρόνο για το τι ακριβώς κάνουν τα διαρθρωτικά ταμεία στα κράτη-μέλη και ένα link με τράπεζα εντομένων όπου έχουμε όλα τα πράγματα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το EMFF. Και θα δείτε λοιπόν εκεί τι ακριβώς ε, γίνεται από το EMFF, ε, το δικό μας το ταμείο, στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η πιο σύντομη απάντηση που ε, θα μπορούσα να δώσω. Όσον αφορά τα στοιχεία, του αριθμούς σχετικά με την εφαρμογή Τώρα, εξαρτάται πώς βλέπει κανείς το ποτήρι, μισοάδιο ή μισογεμάτο. Βεβαίως υπάρχει το γεγονός ότι κατ' ουσίαν έχουμε δαπανίσει το 23% του ταμείου, ε, το 45% είναι δεσμευμένο. Αυτό μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Εγώ προτιμώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μόνο γιατί έχουμε επιτύχει ουσιαστική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά και διότι, όπως είπε και κάποιος ευρωβουλευτής, πρέπει να αναγνωρίσουμε αναγνωρίσουμε τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για να διασφαλίσουν ότι οι ευκαιρίες που προσφέρει το Ταμείο θα τύχουν πραγματικής εκμετάλλευσης. Όσον αφορά την μικρή κλίμακα Σαλία, το Ταμείο, το EMFF, προβλέπει ειδική μεταχείριση για μικρούς αλείς και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ε, ένα ποσοστό 100%. Άρα δηλαδή είναι σαφές ένα μήνυμα ότι εμείς στηρίζουμε ή το Ταμείο στηρίζει τους μικρούς αλείς. Και για τα αμέσως επόμενη περίοδο έχουμε προτείνει να υπάρχει ένα απόθεμα ε, για... Ε, μάλλον να προβλέπονται κάποια μέτρα για μικρού αλεί, ειδικά για αυτού δηλαδή, όταν θα θέλουν να αγοράσουν ένα άλλο σκάφο, ειδικά για αυτού να υπάρχουν ειδικά μέτρα για να καλύπτονται οι ανάγκε του. Και ε, τελικά, όσον αφορά τα SFPAs, Σήμερα το απόγευμα νομίζω ότι θα συζητήσει για πάρα πολλέ από αυτέ τι SFPAs με του συναδέλφου μου. Η προσέγγιση είναι προ τη βιωσιμότητα. Και αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να απαντήσουμε σε ερωτηματικά που υπάρχουν ε, για την βιωσιμότητα των τοπικών ε, στόλων ε, οι συνάδελφοί μου είναι εμπειρογνώμονε. Καλύτερα να τα κουβεντιάσετε μαζί του ε, σήμερα το απόγευμα. Ε, εδώ θα σταματήσω, αλλά αν θέλετε να ρωτήσετε και κάτι άλλο, πολύ ευχαρίστω να σα απαντήσω σε διμερέ επίπεδο ή και κατηδίαν. Πολύ ωραία. Μέχρι την Πέμπτη μπορούν να καταβληθούν, να υποβληθούν με συγχωρείτε οι τροπολογίες. Και αν δεν θέλετε, λοιπόν, δεν χρειάζεται να καταθέσετε ειδική τροπολογία για τον προϋπολογισμό. Ε, επόμενο θέμα είναι η συζήτηση με το Γενικό Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων, που νομίζω ότι είναι παρόν, είναι ήδη παρόν. Άρα, uh, να καλωσορίσουμε τον κύριο Ματζάδο, Γενικό Διευθυντή της Mare. Γνωρίζετε ότι ο Γενικός Διευθυντής ε, είναι εδώ και τέσσερα χρόνια σε αυτή τη θέση. Επίσης θα γνωρίζετε ότι σύντομα θα αποχωρήσει γιατί του ανοίγονται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες και έτσι θα έχει και την ευκαιρία και τη δυνατότητα να περιγράψει τα μεγάλα θέματα και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Σίγουρα κατά τη θητεία σας είχατε και σημαντικές ε, επιτυχίες. Ίσως θα μπορούσατε να σταθείτε και σε κάποιες από τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίζουμε στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Κρίς. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αλίας. Ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερος που με προσκαλέσατε και που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα της αλίας. Τους περισσότερους από εσάς δεν σας γνωρίζω, κάποιους όμως ε, τους θυμάμαι. αρχικά να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για την πολύ δυσάρεστη είδηση που μας ήρθε από τις Αζόρες ότι ο Άντρια Φόρντ, συνάδελφός σας, που θα έπρεπε να είναι εδώ, μέλος αυτής της Επιτροπής, δυστυχώς απεβίωσε και σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν ε, ιδιαίτερα δραστήριος, πολιτικό εκπροσωπούσε την ε, τοπική κοινωνία και σίγουρα θα έχει συμβάλει με πολύ σημαντικό τρόπο ε, στο έργο της Επιτροπής σας. Και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένειά του και τους οικείους του. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, Κρίς, να σε συγχαρώ για την εκλογή σου και να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχεις την αμέριστη υποστήριξη προσωπικά δική μου και της υπηρεσίας μου, όποτε τις ζητήσεις. Και προβλέπουμε σε πολύ στενή συνεργασία για την ε, συνέχιση της ε, χρήσιμης και επικοδομητικής αυτής της συνεργασίας με την Επιτροπή σας. Να καλωσορίσω θερμά και τα νέα μέλη αυτής της Επιτροπής, σε έναν κόσμο θαλασσών και ωκεανών. Η αλληλεία και οι θαλάσσιες υποθέσεις είναι ένα ε, εξαιρετικά ενδιαφέρον ε, και συναρπαστικό θέμα που μας αφορά όλους. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% του πλανήτη μας. Είναι ζωτική σημασίας για την ανθρώπινη ζωή, την ευημερία μας και την ευημερία των επόμενων γενεών. Και σε ό,τι αφορά ε, ε, τα τρόφιμα πολύ υψηλής τροφικής αξίας, αλλά και σε ό,τι αφορά την έρευνα, συγγνώμη, την ενέργεια και άλλους σημαντικούς ε, πόρους. Και σε ό,τι αφορά τον φυσικό κύκλο, αλλά και ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και τεχνολογικής καινοτομίας. Αλλά αποτελεί και μία πηγή έμπνευσης, φαντασίας και ταπεινότητας. Για μεγάλο αριθμό πολιτών, η θάλασσα είναι και κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε παράκτιες περιοχές και 40% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε απόσταση κάτω από 160 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Οι ωκεανοί μας λοιπόν μας ενώνουν Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό για και την ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών. Η Επιτροπή σας παραδοσιακά εστιάζει την προσοχή της στην αλία. Όμως θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα ζητήματα των ωκεανών πιο σφαιρικά και η αλία, η γαλάζια οικονομία και η διακυβέρνηση είναι ζητήματα αλληλένδετα. Και θεωρώ ότι η Επιτροπή σας μπορεί να δραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας τέτοιας ε, σφαιρικής ε, προσέγγισης. Θα ήθελα σήμερα να σας παρουσιάσω τις απόψεις μου για τις βασικές προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες. Φυσικά, με την επιφύλαξη και πιθανών ε, πρωτοβουλειών που μπορεί να αποφασίσει το νέο σώμα επιτρόπων όταν ε, ξεκινήσει τη θητεία του. Κάτι που θεωρώ αυτονόητο είναι ότι οι ωκεανοί σίγουρα θα βρεθούν ψηλά στο πολιτικό θεματολόγιο της επόμενης θητείας. Το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Green Deal είναι η πρώτη και κύρια προτεραιότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίαζε και η νεοεκλεγήσα πρόεδρος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Από τις ευρωεκλογέ είδαμε ότι η διατήρηση του πλανήτη μας και των οικοσυστημάτων μας βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να εισακουστούν λοιπόν αυτές οι ανησυχίες αυτή η πράσινη συμφωνία, το Green Deal, σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει η πρώτη ήπειρος που θα είναι ε, κλιματικά ουδέτερη. Από τους ωκεανούς βλέπουμε τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής, ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, έχουμε μεγαλύτερες ε, καταιγίδε, ε, χάνουμε τους ε, και τη ζωή στους υφάλους και άλλα προβλήματα. Από την άλλη όμως έχουμε και λύσεις γιατί οι ωκεανοί απορροφούν 25% των αερίων του θερμοκηπίου και 90% της πλεονάουσας θερμότητας του πλανήτη. Και για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των ωκεανών μας, για παράδειγμα για την παραγωγή τροφίμων και ενέργειας. Η Πράσινη Συμφωνία αφορά επίσης τη διατήρηση της βιοποικιλότητάς μας. Αυτό περιλαμβάνει την διατήρηση και προστασία θαλασσών και ωκεανών και απαιτεί νέα πρότυπα που θα διέπουν ε, και το εμπόριο και την ε, γεωργία, την αλληλεία και όλα αυτά τα θέματα. Συνολικά λοιπόν σε μια προσπάθεια προστασίας των ωκεανών. Η Πράσινη Συμφωνία αφορά και τα βιώσιμα τρόφιμα σε όλη την αλυσίδα αξιών. Ένας βασικός στόχος της κοινή αλληλευτικής πολιτικής είναι η διασφάλιση της συχνελισιμότητα, ασφάλειας και ποιότητας ε, των προϊόντων ε, που τίθενται σε εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περίπου 60% των ε, θαλασσινών και έτσι είναι μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Θέλει λοιπόν να προωθήσουμε ε, τα βιώσιμα θαλασσινά ως βασικό μοχλό λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση θα αξιοποιήσουμε και τις ιδιωτοκαλλιέργειες. Σημαντικός στόχος είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της ρήπανσης από πλαστικό. Για να μην έχουμε περισσότερα πλαστικά στους ωκεανούς μας τα επόμενα χρόνια από ότι έχουμε ψάρια. Δεν θέλουμε να απορρίπτονται πλέον ε, οι εξοπλισμοί στη θάλασσα που αποτελούν περίπου το 20-25% ε, των απορριμμάτων στους ωκεανούς. Με τη στήριξη της Επιτροπής σας, η Πράσινη Συμφωνία θα γίνει και γαλάζια συμφωνία ή τουλάχιστον θα περιλαμβάνει πολλές αποχρώσεις ε, του γαλάζιου. Θα ήθελα όμως ε, να σταθώ και σε ορισμένα από τα βασικά ζητήματα στα οποία σημειώσαμε από κοινού σημαντική πρόοδο κατά τελευταία πενταετία. Υιοθετήσαμε τέσσερα πολιετή διαχειριστικά σχέδια για τη διαχείριση της αλίας. Ένα για τη Βαλτική, ένα για τη Βόρεια Θάλασσα, ένα για τα δυτικά Ήδατα και ένα για τη Δυτική Μεσόγειο. Το πρώτο πολιετές σχέδιο στη Μεσόγειο που αποτελεί μία νευραλγική θαλάσσια ζώνη. Υιοθετήσαμε και νέους πιο απλούς ε, κανόνες σε ό,τι αφορά την ε, προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Τα λεγόμενα τεχνικά μέτρα. Ο κανονισμός περί τεχνικών μέτρων. Και συμφωνήσαμε επί νέων κανόνων για την βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών μας ε, αλευτικών στόλων και για ένα νέο πλαίσιο συλλογής δεδομένων. Ένα πράγμα είναι σαφέ μετά από όλη αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει. Όταν το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται από κοινού και συμμερίζονται ένα κοινό όραμα, μπορεί να σημειωθεί πραγματική πρόοδο για την διασφάλιση τη ε, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητας ε, τη αλληλεία μα και διατήρηση ε, των θαλασσών και κενών μα μακροπρόθεσμα. Αντιμετωπίζουμε τεράστιες προκλήσεις σήμερα από την κλιματική αλλαγή και το μετριασμό των επιπτώσεων στους ωκεανούς μας μέχρι την καταπολέμηση της απώλειας βιοπικιλότητας στα θαλάσσια οικοσυστήματα, καταπολέμηση της θαλάσσιας ρήπανσης και διατήρηση και προστασία ε, της οικονομικής δραστηριότητα των αλλιών μας και των παράκτιων ε, κοινοτήτων μας. Και βέβαια για την επόμενη θητεία έχουμε πολύ και σημαντική δουλειά να κάνουμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε επί ενός νέου ταμείου θάλασσών και αλίας. Να διασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την επόμενη πραγματική περίοδο που θα ξεκινήσει το 2021. Πρέπει παράλληλα να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα ελέγχου αλίας, το οποίο θεωρούμε ότι πλέον δεν είναι κατάλληλο. Και μέχρι το 2020 πρέπει να φτάσουμε το, την λεγόμενη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δηλαδή τα ετήσια αλλιεύματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τις θάλασσες κάθε χρόνο χωρίς να απλήξουμε τη δυνατότητα του αποθέματος ε, να αναπαραχθεί και να αναπληρωθεί. Και θα πρέπει να αλλοποιήσουμε και την λεγόμενη υποχρέωση εκφόρτωση που θα τεθεί πλήρω σε ισχύ, ε, μάλλον ετέθη σε ισχύ την 1η Πρώτη του 2019. Και έχουμε και την πλήρη απαγόρευση ε, των ε, απορρίψεων ε, αλλιευμάτων στη θάλασσα. Από την άλλη, θα πρέπει να αντιστρέψουμε κατεπηγόντως την ανησυχητική τάση στη Μεσόγειο, όπου υπάρχει τεράστια υπεραλίευση. Είναι η περιοχή του κόσμου που έχει παρουσιάσει τη μεγαλύτερη υπεραλίευση. Τώρα λοιπόν, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ένα κοινό όραμα για τη βιώσιμη αλληλεία. Χρειαζόμαστε περισσότερη και όχι λιγότερη φιλοδοξία. Και θα πρέπει να επανεπιβεβαιώσουμε τον κοινό μας στόχο να έχουμε υγιείς ωκεανούς, να μην αποδυναμωθούν περαιτέρω. Θα σας δώσω ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε έναν από, τους, από αυτούς τους ε, στόχους. Ο κανονισμός ε, της κοινή ελευτικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σαφής. Η μέγιστη βιώσιμη απόδοση θα πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020. Έχουμε σημειώσει πρόοδο σε ό,τι αφορά την επίτευξη αυτού του στόχου τα τελευταία χρόνια σε πολλά τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι σε βρίσκονται στην καλύτερη, στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ. Το 2019 ο αριθμός των ε, τάξ, των ε, ποσοστώσεων που συμβαδίζουν με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση αυξήθηκε σε 59. Αυτό ε, εκπροσωπεί το 78% όλων των ποσοστώσεων που έχουν αξιολογηθεί στα αποθέματα. Και η πίεση προς τα αποθέματα εξεκολουθεί να μειώνεται στον Βόρειο Ατλαντικό. Και έτσι αναπληρώνονται τα αποθέματα. Η βιομάζα είναι κατά 36% αυξημένη σε σχέση με το 2013 στον Ατλαντικό. Από τα δεδομένα λοιπόν βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η βιώσιμη αλληλεία ε, έχει ωφέλη και για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομία. Η βιώσιμη αλληλεία βελτιώνει και τη βιομάζα των αποθεμάτων αλλά συνολικά και την ε, κοινωνική και οικονομική απόδοση του ευρωπαϊκού στόλου. Ένα στόλος που σημειώνει τεράστια κέρδη. 1,3 δις το 2017. Όμως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Ιδίως στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα. Ιδίως ό,τι την κατάσταση των μεσογειακών αποθεμάτων που είναι ιδιαίτερα ενισχυτική. Στη Μεσόγειο λοιπόν περίπου το 87% των αποθεμάτων υπεραλλιεύεται. Φέρουμε συλλογικά την ευθύνη της βελτίωσης της κατάστασης στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να μην κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Όμως ανησυχητική είναι και η κατάσταση τελευταία στη Βαλτική. Όπως ε, υπάρχουν συγκεκριμένα αποθέματα, όπως ο, ο Βακαλάος Ανατολής, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε πολύ ανησυχητική κατάσταση. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στις αλληλευτικές προσπάθειες, αλλά και σε πολλούς άλλους παράγοντες. Και πάλι όμως απαιτείται άμεση ανάληψη δράσης η Επιτροπή σήμερα θα υιοθετήσει κατεπίγοντα μέτρα για την ε, ε, διάσωση των ε, αποθεμάτων της Ανατολικής Βαλτικής από την άμεση κατάρρευσή τους, που θα ήταν καταστροφική για τις παράκτιες κοινότητες της Βαλτικής. Βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει την πρότασή της για τις αλευτικές ε, προσπάθειες και δυνατότητες για το 2020. Τα τάξη λοιπόν, αυτές οι ποσοστώσει ε, θα αποφασιστούν από το Συμβούλιο το φθινόπωρο. Για την Βόρειο Θάλασσα και το Βόρειο Ατλαντικό θα ε, προσδιοριστούν βάσει του ΠΔΛΤΑΠΗ. Η ο βασικό στόχο των προτάσεων τη Επιτροπή θα είναι, όπω είπα, να πετύχουμε την μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα αποθέματα μέχρι το 2020. Αυτό φυσικά θα είναι μια μεγάλη πρόκληση και απαιτεί σημαντικέ και συλλογικέ προσπάθειε από όλου του φορεί. Εάν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να συνεχίσει να είναι παγκόσμιο ηγέτη για τη βιωσιμότητα των ωκεανών, οφείλουμε να εφαρμόσουμε τις δικές μας τις ε, προδιαγραφές και να τηρούμε τις ε, νομικές μας υποχρώσεις ε, στις δικές μας τις θαλάσσιες λεκάνες. Ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίζουμε, μια άλλη πρόκληση, είναι η εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουμε σε μη επιθυμητών αλληλευμάτων. Αυτές οι δεσμεύσεις οφείλουν να οδηγήσουν τον αλλιευτικό τομέα στο να επιλέξει ε, καλύτερα πρότυπα για να υπάρχουν ε, λιγότερα παραλιεύματα. Τον Ιανουάριο του 2019 είπαμε ότι οι δεσμεύσεις αυτές ισχύουν απόλυτα για όλα, όλα τα σκάφη εμπορικής αλίας ε, και ε, για ευρωπαϊκά σκάφη που αλλιεύουν σε ανοιχτή θάλασσα. Όμως πάρα πολλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές ε, προκλήσεις και δυσκολίες στο να εφαρμόζουν αυτές τις υποχρεώσεις. Αυτός λοιπόν ο τομέας είναι πολύ επικριτικός όσον αφορά ακριβώ αυτό το θέμα που έχει σχέση με την κοινή αλλιευτική πολιτική πολλά κράτη-μέλη της προηγούμενης ε, Επιτροπής Αλίας ανοιχτά αμφισβήτησαν αυτή την αρχή ε, της, ε, των δεσμεύσεων για την εκφόρτωση. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη για να τα ενθαρρύνουμε να κάνουν χρήση όλων αυτών των εργαλείων τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την εκφόρτωση και να κάνουν επίσης καλύτερη χρήση των ε, κονδυλίων που υπάρχουν για να εφαρμόζουν ε, καλύτερες τεχνικές και να χρησιμοποιούν πιο επιλεκτικό εξοπλισμό. Εξάλλου ελέγχουμε πολύ προσεκτικά έτσι ώστε όλες ε, οι αιτήσει από τα κράτη-μέλη για εξαιρέσεις από αυτές τις δεσμεύσεις να είναι σωστά αιτιολογημένες και να βασίζονται σε τεκμηριωμένες επιστημονικές συμβουλές. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε οι εξαιρέσεις εγκρίνονται, θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη μορφή κατεξουσιοδότηση πράξεων, οι οποίες κατόπιν ελέγχονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που μπορούν βέβαια να εκφράσουν την αντίρρησή τους. Βεβαίως, ε, είναι απολύτως απαραίτητο και μας απασχολεί το ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι δεσμεύσεις, γιατί υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, ενδείξεις ε, προκύπτουν από ελέγχους που κάνουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν ελέγχουν ικανοποιητικά ε, την ε, εφαρμογή των δεσμεύσεων εκφόρτωσης. Χρειαζόμαστε λοιπόν νέο σύστημα, καινοτόμο σύστημα ελέγχων, όπως διότι αποδείχθηκε ότι οι συμβατικοί έλεγχοι αποδείχτηκαν μη αποτελεσματικοί. Το σύστημα, το ηλεκτρονικό, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εξ αποστάσεως είναι το πιο αποτελεσματικό για να μπορούν τα κράτη-μέλη πράγματι να εφαρμόζουν τις δεσμεύσεις εκφόρτωσης στη θάλασσα. Και γι' αυτό η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση τηλεόρασης ε, κλειστού κυκλώματος, το περίφημο CCTV σύστημα. Αυτό το προτείνουμε στον ε, αναθεωρημένο κανονισμό ελέγχου. Γνωρίζω ότι πολλά κράτη-μέλη κατά, στην προηγούμενη Επιτροπή Ελίας συμπεριλαμβανομένου και του προηγούμενου εισηγητή άσκησαν έντονη κριτική απέναντι σε αυτό το σύστημα κλειστού κυκλώματος ε, πάνω σε αλληλευτικά σκάφη και αυτό το έκαναν κυρίως για λόγους ε, προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η διαφύλαξη αυτών των δεδομένων μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Επιτροπή και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Όμως, η δική μας η πρόταση προβλέπει επίσης ε, ότι ε, τα στοιχεία από το κλειστό αυτό κύκλωμα θα καταγράφονται πάνω στα σκάφη και θα διατίθενται μόνο στους ε, υπαλλήλου του κράτους μέλους ή στους επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν υπάρχει έλεγχος ή κάποια έρευνα. Τα στοιχεία αυτά ε, δεν θα μεταδίδονται ε, σε συνεχή μορφή στις αρμόδιες αρχές ελέγχου του κράτους μέλους. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι σε μία περίοδο όπου κάθε ένας από εμάς ως πολίτης αισθάνεται όταν περπατάει σε ένα ε, μαγαζί ή ε, σταματάει σε ένα βενζινάδικο, εκεί δεν μπορεί να πει τίποτα. Δεν μπορεί να πει ότι ε, δεν θέλω να καταγράφομαι σε κλειστό κύκλωμα ισχύει αυτό και για τα σκάφη, γιατί και τα σκάφη αναπτύσσουν μια οικονομική δραστηριότητα σε ένα χώρο που ανήκει σε όλους μας. Δεν πρόκειται για παραβίαση ε, προσωπικών δεδομένων των αλλιών. Εδώ πρόκειται για το μόνο αποτελεσματικό μέσο που μας επιτρέπει να ελέγχουμε εάν οι κανόνες ε, τους οποίους έχετε αποφασίσει εσείς ε, τα μέλη ε, του Κοινοβουλίου ε, μαζί με το Συμβούλιο αν θέλουμε όλοι αυτοί οι κανόνες να ε, γίνονται σεβαστοί. Εφόσον μιλάμε για τον έλεγχο θέλω να είμαι σαφής και για άλλο ένα πράγμα. Η επιτυχία ή η αποτυχία της κοινή αλληλευτικής πολιτικής εξαρτάται από το κατά πόσον θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική της εφαρμογή ή όχι. Δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την, τα MOUs ε, αν δεν ε, αναθεωρήσουμε το σύστημα ελέγχου. Γιατί το σύστημα αυτό δεν είναι κατάλληλο, καθότι ε, εκφράζει στρατηγικές ελέγχου που είναι απαρχαιωμένες. Είναι τουλάχιστον 10 ετών η πρόταση για την αναθεώρηση αυτού του ελέγχου προβλέπει τον εξυγχρονισμό των ελέγχων, τη χρήση της νέας τεχνολογίας και την ίση μεταχείριση όλων των επιχειρήσεων. Έχουμε προτείνει να μην υπάρχει πλέον χρήση χαρτιού, να εναρμονιστούν τα κριτήρια ε, για ε, σοβαρές παραβάσεις και με τον τρόπο αυτό ο νέος κανονισμός ελέγχου μπορεί να δημιουργήσει ίσες προϋποθέσεις σε όλα τα κράτη-μέλη οποτεδήποτε πρόκειται για την εφαρμογή της κοινή ελληνικής πολιτικής. Τώρα πλέον εναπόκειται σε εσά να δράξετε την ευκαιρία και να εφαρμόσετε ένα φιλόδοξο και σύγχρονο κανονισμό που ε, είναι, κρίνεται ο κατάλληλος και που μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε ε, σωστά την αλληλευτική πολιτική στα ενωσιακά ύδατα. Ε, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση θα προχωρήσει γρήγορα σε αυτή την Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυγχρονίσουμε το σύστημά μας ελέγχου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Και τώρα θα πω λίγα λόγια για την πρόταση της Επιτροπής ε, που αφορά στο EMFF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, αφορά ε, στην περίοδο 20-27. Πρόκειται για το πιο επίγον θέμα που θα κληθείτε να χειριστείτε. Κατά τα τέλη της προηγούμενης θητείας, τον Απρίλη, το προηγούμενο Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση ε, την πρόταση για το EMFF. Μετά από κάποιους μήνες, τον Ιούνιο, ενέκρινε την ε, μερική γενική προσέγγιση. Οι θέσεις ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση. Και υπάρχουν σοβαρές ε, ανησυχίες ε, πρέπει να σας πω από πλευράς Επιτροπής. Γιατί, διότι βλέπουμε ότι αυτά που θέλουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αντιβαίνουν ε, στην δική μας την πρόταση για κοινή ελευτική πολιτική που εγκρίθηκε πριν από έξι μόνο χρόνια. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό το ταμείο, οι συζητήσεις για το EMFF μου προκαλούν μία λύπη ότι είχαμε δεσμευτεί απέναντι στην βιώσιμη ελεία και αυτό εγκαταλείπεται σιγά σιγά. Χάνονται οι κοινοί μας στόχοι. Κατά την άποψή μου είναι απαράδεκτο τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο που τίθεται σε κίνδυνο η κοινή αλληλευτική πολιτική και μάλιστα αντίθετα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς κάποια από τα στοιχεία αν ε, επαναφερθούν στο μελλοντικό IMF, e θα οδηγήσουν ακριβώς εκεί που μόλις τώρα σας παρουσίασα. Θα κάνουμε, φοβάμαι, ένα πολύ επικίνδυνο βήμα προς τα πίσω το οποίο όχι μόνο θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα της αλίας μας, αλλά και θα υπονομεύσει την αξιοπιστία μας σε παγκόσμιο επίπεδο ως ε, πρωταθλητές της βιώσιμης αλίας ε, και υποστηρικτές ε, των στόχων της χιλίτιας. Πλέον εναπόκειται σε εσά στα νέα μέλη της Επιτροπής, αν αυτό πραγματικά επιθυμείτε. Και σύντομα να σας εξηγήσω τις ανησυχίες μας για τρεις ε, πολύ προβληματικές ε, τροπολογίες στην πρώτη ανάγνωση που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν, επενδύσεις ε, σε μικρά αλληλευτικά σκάφη. Αυτό δεν θα μας επέτρεπε να στηρίξουμε νέα σκάφη και την νέα αίρεσιμότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή. Η υποστήριξη για την κατασκευή νέων σκαφών. Αυτό αλλάζει τελείω το στόχο της πρότασης και μπορεί να οδηγήσει σε υπερπλεώνασμα Και αυτό ε, θα επηρέαζε αρνητικά την ε, βιώσιμη αλία. Δεύτερον, η, τα επιδόματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφήγηση σκαφών ε, Αυτά έκλεισαν το 2004. Ξέρετε γιατί, διότι οδήγησαν σε μια κατάσταση όπου είχαμε υπερπλεόνασμα στον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αλληλευτικό σκόλο, στόλο. Και που είχε οδηγήσει αυτό, είχαμε και ως αποτέλεσμα υπεραλήψη πολλών αλληλευμάτων. Τώρα, αν επανέλθουν τέτοιου είδους επιδόματα, αυτό αντιβαίνει, όπως σας είπα, στην πολιτική, την κοινή που αποφασίσαμε το 2013 και μόνο αυτό, αλλά έτσι θα ε, παραβιάζουμε και τις ε, υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει ε, στο πλαίσιο των στόχων της χιλιετίας. Και επιπλέον θα, τεθούν, ε, θα τεθεί σε κίνδυνο η θέση που έχουμε καταλάβει ε, στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τον ΠΟΕ. Και επιπλέον ε, θα απέκλειε την συγκέντρωση κονδυλίων για άλλους πολλούς ε, σημαντικούς στόχους, όπως είναι η βελτίωση της επιλεξιμότητας και η βελτίωση των ε, προϋποθέσεων, να υπάρχουν ίσες προϋποθέσεις ανταγωνισμού σε πολλά κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου, το EMFF ε, ίσως να οδηγήσει σε κάποιες αποτυχίες, αλλά δεν θα επαναφέρει επιδόματα κυρίως σε τομείς όπου τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κέρδη ρεκόρ. Η επαναφορά των επιδομάτων θα οδηγήσει σε σημαντική στρέβλωση της αγοράς. Θέλω λοιπόν να είμαι απόλυτα σαφής. Να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση όσον αφορά τη θέση της Επιτροπής. Εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχουν επιδόματα τα οποία βελτιώνουν τις ε, συνθήκες εργασίας στα σκάφη. Είμαστε υπέρ του να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις που προάγουν την ασφάλεια ε, πάνω στα σκάφη. Αλλά όλα αυτά μπορούν να γίνουν χωρίς να αυξηθεί ο αριθμός των ε, σκαφών. Γιατί να χρειάζονται επενδύσεις να, αναφυγηθούν νέα σκάφη. Ε, το τρίτο που μας ανησυχεί είναι η διαγραφή της εισφοράς του 30% του MFF ε, σε στόχους ε, κλιματικούς. με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχουν κάποιες οριζόντιες δράσεις που προβλέπονται για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε σε κάποιες αλλαγές που ζήτησε το Κοινοβούλιο και αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στην απάντησή μας που ε, είναι στη διάθεσή σας σε όλες τις γλώσσες. Οι υπηρεσίε μου και εγώ προφανώς και είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε και άλλες εξηγήσεις ε, πριν ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι κατά τη διάρκεια των επικείμενων τριμερών διαλόγων τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο θα κληθούν να αποφασίσουν κατά πόσον παραμένουν στο στόχο τους που είναι βιώσιμη αλία ή όχι κατά πόσον θέλουν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες της επόμενης γενιάς, κατά πόσον επιθυμούν να προχωρήσουν προς τα εμπρός ή να οπισθοδρομήσουν προς τα πίσω, αν θέλουν το μακροπρόθεσμο ή το βραχυπρόθεσμο. Ε, πριν από κάποιες εβδομάδες ε, οι περισσότερες πολιτικές ομάδες ζήτησαν η βιωσιμότητα να είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες για την νέα Επιτροπή η πρόεδρος της Επιτροπής που εξελέγει, ακούσαμε ότι θεωρεί τη βιωσιμότητα προτεραιότητα και ισχύει αυτό και για σας, τα μέλη της Επιτροπής. Αξιότιμοι βουλευτές. Ε, και πριν ολοκληρώσω θέλω να πω και δύο μόνο πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι η μεγαλύτερη αλληλευτική και θαλάσσια δύναμη και όπως σας είπα η μεγαλύτερη ε, κοινή αγορά για αλληλευτικά προϊόντα στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είναι ευθύνη μας να βελτιωθούν οι προδιαγραφές βιωσιμότητα σε διεθνές επίπεδο και ε, να παραμείνουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες ασφαλείς, καθαροί, όχι μόνο μέσα στα δικά μας σύνορα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε παγκόσμιες προκλήσεις και παράλληλα να διασφαλίσουμε ίσες ε, προϋποθέσεις ε, για τους ε, εμπορευόμενους. Τα προβλήματα στη θάλασσα είναι διασυνοριακά. Είναι σημαντικό το τι θα κάνουμε για να ενισχύσουμε τους πολυμερείς κανόνες. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να δράσουμε σε όλα τα επίπεδα, το ενωσιακό, το περιφερειακό, αλλά και το διεθνές επίπεδο. Τα βασικά μας εργαλεία για να προάγουμε την βιώσιμη αλληλεία και την καλύτερη διαχείριση είναι η δουλειά στους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή φόρα και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών η δουλειά σε περιφερειακούς οργανισμούς διαχείρισης αλίας, οι διμερείς και πολυμερείς αλλιευτικές συμφωνίες, η διεθνής μας πολιτική και η πολιτική μας για την αντιμετώπιση ε, παράνομης ε, και μη καταγραφόμενης ε, ε, αλίας, IOU όπως είναι γνωστή. Εμείς ε, παρακολουθούμε ε, από πολύ κοντά τις συμφωνίες. Οι συνάδελφοί μου από τη δική μου την υπηρεσία σήμερα το απόγευμα θα έρθουν στην Επιτροπή σας για να μιλήσετε ήδη για κάποια από αυτά τα θέματα. Η πολιτική αλίας αυτό σημαίνει ότι καλούμεθα και να έχουμε μια βιώσιμη μπλε οικονομία. Χωρίς την βιώσιμη μπλε οικονομία δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε ενωσιακές εταιρείε να επωφεληθούν από μια δυναμική οικονομία των ωκεανών που θα σέβεται πλήρως ε, κοινωνικές ε, και περιβαλλοντικές ισορροπίες. Η αξία της ε, γαλάζιας οικονομίας προβλέπεται ότι θα διπλασιαστεί την επόμενη δεκαετία, θα φτάσει μέχρι το 2030 το 1-3. Μιλάμε το διπλάσιο ΑΕΠ σε αναδιόμενους ε, τομείς ε, σε πάρα πολλούς που μεταξύ αυτών αναφέρεται και η μπλε βιοτεχνολογία. Όλα αυτά θα αλλάξουν και θα διαφοροποιήσουν την ε, θαλάσσια οικονομία. Ελπίζω να συνεργαστούμε και με αυτή την Επιτροπή έτσι ώστε να δημιουργηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθούν να λειτουργήσουν οι ε, φορείς ε, για να ε, ευημερίσουν στην ευρύτερη οικονομία των ωκεανών. Αξιότιμα μέλη, πριν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να πω λίγα μονολόγια για το Brexit. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Επιτροπή συνεχίζει να δουλεύεται πάνω στην παραδοχή ότι θα υπάρξει μια συντεταγμένη αποχώρηση ε, με βάση τη συμφωνία αποχώρησης που προβλέπει μια μεταβατική περίοδο και προβλέπει και διμερείς ε, διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε μια μακροχρόνια συμφωνία για τις οικονομικές μας σχέσεις και μετά το 2020. Μετά λοιπόν τη μεταβατική περίοδο και όσον αφορά τη μακροχρόνια σχέση μας με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο βασικός μας στόχος ε, θα είναι να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη χρήση των πάνω από 100 αλληλευτικών αποθεμάτων ε, που από τη μια μέρα στην άλλη ε, θα τα μοιραζόμαστε με το Μενωμένο Βασίλειο επί τη βάση διαπραγματεύσεων ε, που θα ακολουθήσουν με βάση τις οδηγίες που χαράχτηκαν το 2018. Αυτό είναι όλο πάρα πολύ δύσκολο με την ε, Νορβηγία έχουμε 7 αποθέματα. Ήδη εκεί οι διαπραγματεύσει είναι πάρα πολύ δύσκολε ε, κάθε χρόνο. Τώρα με το Ηνωμένο Βασίλειο από τη μια μέρα στην άλλη ε, θα κληθούμε να διαχειριστούμε 100 αλληλευτικά αποθέματα κοινά επί των οποίων θα πρέπει να έχουμε διαπραγματεύσεις. Όμως έχει αυξηθεί περισσότερο τους τελευταίους μήνες ο κίνδυνος του να μην υπάρξει τελικά συμφωνία. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, προετοιμαστεί πολύ καλά και για το ενδεχόμενο του αποκαλούμενου σκληρού Brexit. Ειλικρινά ελπίζω ότι αν τελικά υπάρξει Brexit, παρόλα αυτά θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχημένες αλληλευτικές μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και πέρα από την ημερομηνία αποχώρησης. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ευκαιρία που μου δώσατε να έχουμε σήμερα αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Και προσβλέπω ε, στο να απαντήσω σε ερωτήσεις που ίσως έχετε. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε να έχετε έτσι μια σφαιρική εικόνα της κατάστασης και παρόλα αυτά δεν μπήκα και σε άλλα θέματα που θα εξεταστούν περισσότερο σήμερα το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, ε, όπως σας είπα, είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω ενδεχομένως σε ερωτήσεις. Και πάλι λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή που θα συνεργαστούμε προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μασάδο. Μας θυμήσατε πολλά σημαντικά πράγματα, ότι το 87% είπατε, δηλαδή κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη στην Αλία και εσεί ω Κομισιόν πρέπει να αναρωτηθείτε κατά πόσον παρά τι ε, νομοθετικέ διατάξει που έχετε εισαγάγει αντιμετωπίζετε την κατάσταση. Και πριν στραφώ στα μέλη, για το EMFF είπατε ότι οι τροπολογίες που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο δημιουργούν μια κατάσταση κατά την οποία ε, υποσκάπτουμε τους στόχους βιωσιμότητα για την αλληλεία. Αλλά μην περιμένετε το κοινοβούλιο να αλλάξει τη θέση του, γιατί θεσμικά υπερασπιζόμαστε μια θέση που είχε υιοθετηθεί σε πρώτη ανάγνωση. Θα έχουμε αυτήν την αντολή διαπραγμάτευση ε, για το Συμβούλιο. Μπορεί να μην μας αρέσει ούτε εμάς ούτε εσάς. Αν θέλετε να ξαναδείτε την πρόταση, από εσά εξαρτάται. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται σε αυτήν την τοποθέτηση. Δηλαδή, αν συμφωνείτε, μην αποφεύγετε την πραγματικότητα. Εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε πράγματα τόσο ουσιαστικά όσο εσείς που την έχετε αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, έχουμε περί τη μία ώρα, ναι, συναδελφοί, μπορώ να εκφράσω και τη δική μου άποψη και την ίδια στιγμή να υπερασπίζομαι και τη θέση του Κοινοβουλίου, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε, όπως έλεγα, μία ώρα. Δεν θα ήθελα Ομάδε ερωτήσεων και απαντήσεων. Θα ήθελα σύντομε ερωτήσει και απαντήσει από τον ε, Γενικό Διευθυντή. Ξεκινούμε από του συντονιστέ θεωρητικά μέχρι τα τρία λεπτά. Αν μπορείτε πιο σύντομα θα σα ήμουν ευγνώμων και ένα λεπτό για του υπόλοιπου. Ο κύριο Μιανμόν, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ ε, τον κύριο Μασάδο για την παρουσία του, ευχαριστώ για την ε, προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια απέναντι σε στόχους και καθήκοντα πολύ σημαντικά και όχι μόνο στις Βρυξέλλες πλέον. Για τη νέα λοιπόν ε, Κομισιόν θα ήθελα να ελπίζω ότι θα γνωρίζει όχι μόνο τα θέματα περιβαλλοντικά και της βοησιμότητας που συμφωνούμε, αλλά και τη σημαντική οικονομική και κοινωνική διάσταση της πολιτικής αλίας. Και η Επιτροπή Αλίας δεν μπορεί να ξεχάσει κάτι τέτοιο. Έχουμε άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στον τομέα αυτό στη μεταποίηση, στην ίδια την αλληλεία, σε πολλά συνδεδεμένα επαγγέλματα. Τώρα αναφερθήκατε σε αυτούς τους ε, μήνες ε, ε, και τα επόμενα χρόνια, ξεκινώντας και τη νέα θητεία, μιλούμε για το Ταμείο. Σε αυτό το, στο πλαίσιο αυτού του περίπλοκου φακέλου δεν θέλω να τοποθετηθώ από τις ουσίες, αλλά γνωρίζουμε ότι η, η έκθεση του οίκου αυτού ε, υιοθετήθηκε σε πρώτη ανάγνωση με ευρύτατη η πλειοψηφία. Ε, η Κομισιόν μπορεί να έχει κάποιες προτιμήσεις, αλλά γι' αυτό έχουμε τριμερείς διαλόγους. Για να βρίσκουμε, να διερευνούμε συνένεση και συνεννόηση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει κανείς να πλήξει τις διεθνείς δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Αλίας. Και δεν είναι θέμα αλλιευτικής δυνατότητας. Είναι θέμα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των σκαφών. Και είναι πολύ σημαντικό για την ανανέωση των αλλιέων των ίδιων. Αλλιώς δεν θα επιτύχουμε ανανέωση χωρίς να μπορούμε να φροντίσουμε τα σκάφη. Είχαμε προ πρόσφατα ε, ένα ρεπορτάζ στην Ισπανικό Τίμο για την Παγιώνα, θα το γνωρίζετε ως Πορτογάλος που είστε, ότι δεν, έχουν, δεν έχουμε πια ψαράδες στο χωριό. Έχουν εγκαταλείψει το χωριό. Δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα κάποιο επίπεδο ε, ποιότητα ζωής για τους αλληλείς και τις οικογένειές τους και τις ζώνες των πληθυσμών που κατοικούν σε περιοχές που εξαρτώνται από την ε, οικονομική αυτή δραστηριότητα. Είχαμε φτάσει και στο παρελθόν σε διάφορες περιπτώσεις σε συμφωνίες, σε τριμερείς διαλόγους και ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι και πάλι θα φτάσουμε σε ισορροπημένη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ερωτήσεις ε, απτέ. Πολύ σύντομα. Ε, Υποχρεώσει εκφόρτωση. Τι κόστο έχουμε για τι επιχειρήσει. Δεύτερον, τι προετοιμάζουμε για πιο μετά μια νέα μετά το 29 κοινή πολιτική. Επίσης, στον βορρά της Μαυριτανίας έχουμε μπλοκάζ, κάθε δύο εβδομάδες ε, έχουμε νέο πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που εκπροσωπώ ε, εκπροσωπούν μεγάλη ανησυχία για αυτές τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Η MFF, λέει ο Πρόεδρος, υποχρεώσεις εκφόρτωσης, Μαυριτανία, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτηση, λέει ο κύριος Μασάδο. Γνωρίζω ότι υιοθέτησε μια πρόταση σε πρώτη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή αυτή έχει πάρα πολλά νέα μέλη και είναι καλό να καταστήσουμε σαφής ποια είναι η ανησυχία της Κομισιόν, την οποία βεβαίως είχαμε εκφράσει κατά διάρκεια των τριμερών διαλόγων είναι καθήκον μου βεβαίως να έρθω εδώ και να εκφράζω την θέση επί της οποίας η Κομισιόν έχει κάποιες ανησυχίες και από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε πώς θέλετε να προσεγγίσετε τους τριμερείς διαλόγους για τις υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Αυτές προϋποθέτουν οι αλληλείς να αλλάξουν τον τρόπο που αλλήλευαν στο παρελθόν να έχουν πιο επιλεκτικό εξοπλισμό, να έχουν διαφορετικές τεχνικές μεθόδους αλίευσης και αυτό απαιτεί μια προσπάθεια και οπωσδήποτε ένα κόστος προσαρμογής. Όμως, οι υποχρεώσει εκφόρτωση είχαν συμφωνηθεί από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και υποθέτω ότι επιθυμείτε ως Κοινοβούλιο να εκτελέσουμε, να υλοποιήσουμε αυτά που αποφασίσατε και συνομοθετήσατε. Εδώ και δύο χρόνια και άνω συζητούμε πράγματα με τα κράτη-μέλη. Τη χρήση των διαφορετικών ε, μέσων πολιτικής που είναι διαθέσιμα υπό την κοινή πολιτική αλίας. Τη χρήση ταμείων κονδυλίων του MFF. Και πρέπει να σας πω ότι δεν χρησιμοποιούνται και τόσο πολύ, δεν απορροφώνται τόσο καλά τα διαθέσιμα κονδύλια δεν λέω ότι όλα αυτά είναι εύκολα, είναι δύσκολα, συμφωνούμε, αλλά δεν θέλουμε η πολιτική αυτή που συναποφασίστηκε από εσάς και το Συμβούλιο το 2013 να μείνει στο περιθώριο, να μείνει εκτός και να έχουμε τις απορρίψεις στη θάλασσα, να συνεχιστεί αυτή η τακτική. Εάν θέλουμε να ελέγξουμε το φαινόμενο αυτό, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω CCTV δεν μπορούμε να ελέγξουμε χωρίς κάμερα, με αέριους ελέγχους κτλ. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες σχετικά με αυτό. Και βεβαίως ήταν αντιφατικό αυτό το θέμα της χρησιμοποίησης των κλειστών κυκλωμάτων των τηλεοπτικών πάνω στα σκάφη, αλλά πρέπει να σας πω ότι και οι οδηγοί των ε, φορτηγών έχουν συστήματα που επιτηρούν πότε οδηγούν, πότε κοιμούνται, ε, με τι ταχύτητα πηγαίνουν κτλ. χρειαζόμαστε CCTV τουλάχιστον εκεί που φορτώνονται τα, ψάρια. Αν θέλετε υλοποίηση, χρειαζόμαστε μέσα ελέγχου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η, νέα ΚΑΠ μετά το 2021. Ο κανονισμός ΚΑΠ ε, προβλέπει ότι μέχρι το τέλος του 2022 η Κομισιόν θα υποβάλει σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έκθεση για την υλοποίηση της ΚΑΠ. Και μετά την συζήτηση της έκθεσης αυτής θα πρέπει να δούμε πρέπει να, μετα... να μεταρρυθμιστεί προς ποια κατεύθυνση, πότε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτά θα συμβούν κάπως αργότερα εντός της θητείας της δικής σας. Και εδώ έχουμε πολύ, δύο πολύ σημαντικά συζήτημα. Η πλήρης υλοποίηση και δεύτερον το να χειριστούμε το Brexit που θα έχει αντίκτυπο επί της ΚΑΠ. Και όταν θα έχουμε δύο αυτά τα δύο, τότε θα είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι για να δούμε πώς μπορούμε να πάμε προς τα εμπρός. Το θέμα της Μαυριτανίας την περασμένη εβδομάδα είχε ήδη τεθεί. Οι συνάδελφοι στην Χαβάτε ε, ε, συζήτησαν με τις Μαυριτανικές Αρχές και πάλι αυτή την εβδομάδα θα είναι εκεί οι συνάδελφοι. Προσπαθούμε να βρούμε λύση, αλλά μέχρι στιγμή ε, διεξάγεται μια συζήτηση μεταξύ αρχών σε συγκεκριμένε κυβερνήσει. Η κυρία Αγγιλάρ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Ματσάδο. Και πάλι. Καταρχά, η κρίση στη Μαυριτανία είναι πολύ σημαντικό θέμα. δύσκολο να βρεθεί καλή λύση, αλλά έχει πάυσει η μια εβδομάδα, οκτώ μέρες θεωρά, πρέπει να βρούμε λύση. Μας είπατε ότι οι συνάδελφοι ασχολούνται, αλλά είναι άμεση ανάγκη η λύση. Για το Brexit ήθελα να καταλάβω κατά πόσον η υπηρεσία σας εργάζεται ε, εν ώψη της προθεσμίας 31 Οκτωβρίου δεν, από ό,τι εμείς καταλαβαίνουμε τα πράγματα δεν έχουμε καλά σημάδια τέλος πάντων αλλά ήθελα να καταλάβω εάν πέραν μιας συμφωνίας για την αλία μπορούμε να έχουμε κάτι άλλο κάτι περισσότερο εάν έχετε προχωρήσει στην υπηρεσία σας για το θέμα αυτό για το Μαρόκο ε, πολύ χαιρόμαστε που ο Ισπανικός στόλος ε, σημαντική παρουσία εκεί έχει επανέλθει στο Μαρόκο και για το Βιετνάμ θα έχουμε μία έκθεση για την ε, συμφωνία την εμπορική αλλά ήθελα να σας πω το εξής έχει κίτρινη κάρτα το Βιετνάμ στην Αλία ήθελα να καταλάβω ποια είναι η άποψη της Κομισιόν για την συμφωνία αυτή πέρα από τα λοιπά εμπορικά ζητήματα επί των οποίων δεν θα τοποθετηθώ η σύσταση μιας ε, εμπορικής συμφωνίας με μια χώρα η οποία έχει παράνομη στάση στην ε, θέματα της αλληλείας ε, γιατί θα ήταν πολύ σημαντικό και για την Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων. Για την ιδεατοκαλλιέργεια αναφερθήκατε πολύ σύντομα. Είναι αλήθεια ότι είναι πολλά τα θέματα και λίγος ο χρόνος, αλλά η ιδεατοκαλλιέργεια στην Ευρώπη χρειάζεται μια υποστήριξη. Γιατί πάμε προς τα πίσω. Δεν κινούμαστε προς τα εμπρός έχουμε άλλες χώρες στον κόσμο με πολύ πιο συγκεκριμένη και στοχευμένη κατεύθυνση που προχωρούν προς τα εμπρός. Εμείς ε, φοβούμε πως ε, κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Θα χρειαζόμασταν υποστήριξη για την υδατοκαλλιέργεια γενικώ τα επόμενα χρόνια. Και κλείνω ε, ε λέγοντας ότι προκαλείται λίγο με το IMFF. E με την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Ε, Σα σέβομαι πολύ, δεν θέλω να πω άλλα. Τώρα δεν θέλω δηλαδή να υιοθετήσω μια πιο επιθετική στάση, αλλά υπήρξατε προκλητικός με αυτά που είπατε. Εδώ υιοθετήθηκε μια γνωμοδότηση με σαφή πλειοψηφία. Ε, υπάρχουν διάφορες απόψεις, αλλά θα σας πω το εξής. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Ένα από τα προβλήματα της χαμηλής απορρόφησης σήμερα είναι ο τρόπος που έγινε. Πρέπει να πω. Ναι, τα επιχειρησιακά προγράμματα ε, εγκρίθηκαν πολύ αργά. Κλείνω, Πρόεδρε. Αλλά στο EMFF ελήφθησαν αποφάσεις και μέτρα που ήταν αδύνατον να εκτελεστούν. Ελπίζω να έχουμε κάποια άλλη δυνατότητα πλέον. Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε, που μακρηγόρησα. Σα ευχαριστώ. Θα, συζητήσουμε το απόγευμα το Βιετνάμ λεπτομερέστερα, λέει ο πρόεδρο. αλλά είναι σημαντικό ότι αν θέλουμε να σταματήσουμε, να περιορίσουμε την ε, παράνομη αλλήλεια, είναι σημείο κλειδί είναι η διαπραγμάτευση ε, η Συμφωνία Ελευθέρωση αλλαγών. Δεν ξέρω καν γιατί προχωρούμε, ενώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Ε, σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε για το Brexit και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Αγγιλάρ για το Brexit. Ναι, οι υπηρεσίες μας εργάζονται ήδη για μελλοντική συμφωνία. Το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα συζητήσει στο Συμβούλιο. Θα υπάρξει εντολή προς την Κομισιόν, αλλά η προετοιμασία έχει γίνει. Και εργαζόμαστε σε αυτό συστηματικά. Γνωρίζουμε απολύτως καλά ποιο είναι το πρόβλημα, ποιε είναι οι προκλήσει και ποια είναι η κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Η κίτρινη κάρτα, το Βιετνάμ και η επικύρωση της ε, συμφωνίας πράγματι ήταν ένας μοχλός αυτό ώστε να του κάνουμε να αλλάξουν τη στάση τους, την πολιτική τους. Η συμφωνία διαπραγματεύτηκε και τώρα κλείσαμε και τώρα μπροστά μας έχουμε την επικύρωση. Αυτό που πρέπει να δει κανείς και θα είμαι πολύ σαφής είναι ότι οι αλλαγές που απαιτούνται για να καταπολεμήσει κανείς την παράνομη λαθρεία και έναρχη αλεία στο Βιετνάμ και να πάμε σε πιο βιώσιμη αλεία θα σημαίνει υιοθέτηση νομοθεσίας, υιοθέτηση συστημάτων ελέγχου, περισσότερο προσωπικό. Στην περίπτωση της Ταϊλάνδης αυτό χρειάστηκε 3,5 χρόνια στην περίπτωση της Ταϊβάν επίσης, 3,5 χρόνια πρωτού άρουμε την κίτρινη κάρτα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μοχλό της μη επικύρωσης για τρία χρόνια, γιατί θα χρειαστεί χρόνος. Δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα έλεγα όμως επίσης, ακόμα και αν επικυρωθεί η συμφωνία αυτή, δεν μας εμποδίζει τίποτα, εφόσον δεν κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και εφόσον ε, εφόσον υπάρξει απαραίτητο να πάμε σε κόκκινη κόρτα, δεν μας εμποδίζει τίποτα να κλείσουμε και υφισταμένης της FTA την αγορά μας σε προϊόντα αλληλείας από το Βιετνάμ. Δηλαδή εγώ έτσι θα το έθετα. Νομίζω ότι είναι μια τέλος πάντων ισορροπημένη εικόνα αυτή που σας δίνω. Για την υδατοκαλλιέργεια συμφωνώ απολύτως μαζί σας αναπτύσσεται και πάλι στην Ευρώπη, αλλά πολύ βραδύτερα από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου. Μερικά από τα προβλήματα που είχαμε με τον τομέα αυτών είναι τα διηγητικά, η αδειοδότηση. Σε κάποια κράτη-μέλη χρειαζόταν πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια για να πάρει άδεια. Γιατί πήγαινε μεταξύ διαφορετικών υπουργείων, γραμματιών, ε, ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ζώνη τάδε για υδατοκαλλιέργεια κτλ. Δηλαδή ένα επενδυτή, αν θέλει πρώτα πέντε χρόνια για την άδεια, μετά θέλει άλλα τρία για να έχει επιστροφή στην επένδυσή του, κανείς δεν στρέφεται σε αυτό. Εμείς τώρα θα επανεξετάσουμε λοιπόν τις κατευθείαν γραμμές για την υδατοκαλλιέργεια στην Ένωση, ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα. Αντιλαμβανόμαστε, γνωρίζουμε πλήρως και πιέζουμε τον κλάδο, μάλλον πιέζουμε το πλαίσιο να απλουστεύσει τις διοικητικές διαδικασίες για τις, επιχει... επιχειρήσεις. Ήμουν προκλητικός για το IMFF. E ναι, μερικές φορές είναι και χρήσιμο να είσαι λίγο προκλητικός, αλλά δεν ήμουν και τελείως προκλητικός. Όταν βλέπω κάποια κράτη-μέλη να ζητούν να επανεισαγάγομαι επενδύσεις για την ε, κατασκευή καφών μέχρι 40 μέτρα, τότε το προκλητικό δεν είναι καν επίθετο που να μπορεί να καλύψει το φαινόμενο. 40 μέτρα. Γνωρίζω ότι στο λιμάνι του Βίγκο ε, κατασκευάζονται 35 σκάφη και το τελευταίο έτος 5 καινούρια με ιδιωτικού πόρους. Δηλαδή δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή επένδυση και χρηματοδότηση, εφόσον έχουμε ιδιωτικούς πόρους, αλλά ναι, υπήρξα λίγο προκλητικός και πιστεύω ότι θα βρούμε κοινό έδαφος μέσω των τριμερών διαλόγων. Να δεν έχουμε και πολλή ώρα. Να το έχετε αυτό κατά νου. Κύριο Σκάλσκι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναφερθήκατε σε πολλά ζητήματα ε, και θα έρθουμε αντιμέτωποι με πραγματικές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Μιλήσατε για το Brexit, μιλήσατε για τους ωκεανούς εν γέννη και το θέμα της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής. Ε, σίγουρα και η επίτευξη των στόχων της κοινή ελευθερικής πολιτικής θα μας απασχολήσει, η υλοποίησή της, αλλά και ενδεχομένω η μεταρρύθμισή τη, εάν ε, οι αξιολογήσεις δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Η υλοποίηση λοιπόν τη ελευθερικής πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τι περιβαλλοντικέ και κλιματικέ προκλήσει ε, σε ό,τι αφορά την προστασία τη βιοποικιλότητα, αλλά ε, και για να αποφέρει καρπού αυτή η πολιτική για στόχους, για κλάδους μάλλον που απασχολούν πολλούς, δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας και υποστηρίζει τις κοινότητες από τις οποίες προερχόμαστε πολύ. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε και με την επιστηστική ασφάλεια της υπήρου μας. Όλα αυτά μας απασχολούν όταν μιλούμε για την αλληλεία και την ιδετοκαλλιεργία. Υπάρχει και το ε, έτθα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεδομένο των προκλήσεων, να υπάρχει δηλαδή ένας φιλόδοξος προπολογισμό. Εμείς θέλουμε ε, αύξηση προλογισμού σε σχέση με τις προτάσεις που έχουμε ακούσει. Επίσης, διακύβευμα είναι να εκτελεστεί αυτός ο προπολογισμός και πραγματικά να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του κλάδου, όπως για παράδειγμα το να έχουμε πιο καθαρά, πιο ασφαλή, πιο επιλεκτικά σκάφη. Ο κλάδος δεσμεύεται προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να υποστηρίξει το Ταμείο αυτή την προσπάθεια. Αντίστοιχα, θα πρέπει να δεσμευτούμε και να, να ικανοποιήσουμε τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω. Και αν θεωρούμε ότι αυτές οι επιδοτήσεις ε, είναι επιζήμιες, πρέπει εμείς να θέσουμε το ερώτημα και κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων να ε, θίξουμε αυτό το ζήτημα και να ε, διασκεδάσουμε τις ε, ανησυχίε. Συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε, λέει ο Πρόεδρο, αλλά παρακαλώ προχωρήστε προ το ερώτημα. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πολύ απλό το ερώτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να υποστηρίξει μια αύξηση του υπερπολογισμού του ΕΤΘΑ όπως επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά ένα ερώτημα για τον Brexit, παρότι δώσατε κάποιες απαντήσεις. Είναι απλό το ερώτημα. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία θα κινηθείτε όσο γίνεται πιο γρήγορα για μια αλληλευτική συμφωνία. Και τρίτον, όλοι γνωρίζουμε για την κλιματική αλλαγή και για την βιοπικιλότητα ότι έχουμε περίπου μια δεκαετία για να ανταποκριθούμε και να αντιδράσουμε. Από τα, τη δεκαετία, τα πέντε χρόνια θα καλύψει η τρέχουσα θητεία. Ποια θα είναι λοιπόν τα μέτρα που θα πάρετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν θα αυξήσει η Επιτροπή τον προπολογισμό. Γνωρίζετε την πρόταση της Κομισιόν, η οποία αφορά μία μείωση σε ονομαστικούς όρους της τάξης του 5% ε, που έχει να κάνει με την ε, αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι το σύστημα που έχει υιοθετηθεί για, υιοθετηθεί για όλα τα ταμεία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αφού αποχωρεί ένα κράτος μέλος, ε, μειώνονται και τα κονδύλια που έχουμε να διαθέσουμε στα κράτη-μέλη. Δεν σημαίνει ότι μειώνουμε δηλαδή από και πέρα τα κονδύλια του ΕΤΘΑ. Δεύτερον, για το Brexit. Ναι, βεβαίως. Ε, αν υπάρξει αποχώρηση χωρίς συμφωνία, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη διαπραγμάτευση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως θέλει δύο η διαπραγμάτευση. Δεν φτάνει να λέμε εμείς ότι θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως, από πλευρά Κομισιόν, εμείς είμαστε απολύτως έτοιμοι και απολύτως διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να έχουμε αλληλευτική συμφωνία των συντομότερων δυνατών. Τώρα, για την αλληλευτική και θαλάσσια πολιτική που είπατε, πρέπει πρώτα να χωνέψουμε εντό αγωγικών τον αντίκτυπο του Brexit στην αλληλευτική πολιτική μας. Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσουμε την υλοποίηση της πολιτικής μας και μέσα στα επόμενα χρόνια να επανέλθουμε στα τέλη του 2022 στο Κοινοβούλιο με μια έκθεση για την ε, υλοποίηση της ελευθερικής πολιτικής για να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να δούμε τι θα γίνει με τον Brexit και μετά να δούμε ποιες θα είναι, ποιες θα είναι οι απαραίτητες προσαρμογές. Σε Thank you, Ευχαριστώ. Um, Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο θέμα των επιδοτήσεων, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προστατεύσουμε ή για να λελατίσουμε τους ωκεανούς και τα αποθέματα. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις ε, της αλίας. και για την υπερβολική ικανότητα και την υπεραλίευση. και τις επιδοτήσεις που συμβάλλουν στην παράνομη λαθρέα και άναρχη Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει επίσης μια διεθνή συμφωνία για, την, για τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναφέρεται. Ο 14-6, λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, απαγορεύει τις επιδοτήσεις που μπορούν να βλάψουν την ε, αλευτικούς πόρου μέχρι το 2020. Όμω βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ρωτώ λοιπόν κύριε Ματσάδο, πώς μπορείτε να μας ε, διαβεβαιώσετε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα δοθούν επιδοτήσεις που θα στηρίζουν τη βιώσιμη αλία, τις βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Αλλά αυτό θα γίνεται με τρόπο το ώστε να μην αντιβαίνει στα όσα λέμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αυτά που λέμε και εκτός να τα ελοποιούμε και εντός. Να μην ε, φανούμε λοιπόν ως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση των Αντιφάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Σάλβαν. Οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη, στο θεματολόγιο του 2030 δηλαδή, δεν προσυπογράφει μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και από όλου του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων του ΟΗΕ. Μεταξύ αυτών και των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών των στόχων έχουμε και τον ε, στόχο 14, η ζωή στη θάλασσα που αναφέρατε κι εσείς. Και εκεί ένας από τους στόχους είναι μέχρι το 2020 του χρόνου να ολοκληρωθεί μια διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του ΠΟΕ που θα απαγορεύει τις επιζήμιες επιδοτήσεις που οδηγούν σε υπεραλίευση και τις επιδοτήσεις που προωθούν την παράνομη λαθρέα και ε, άναρχη αλία. Αν χάσουμε αυτή την προθεσμία του 2020, θεωρώ ότι αυτό θα διακινδυνεύσει ε, την αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Δεύτερον, άλλοι εταίροι στη Γενέβη ανησυχούν ιδιαίτερα με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι της Κομισιόν, που ετέθησε στο τραπέζι του ΠΟΕ πριν από δύο χρόνια ήταν η απαγόρευση των επιδοτήσεων που οδηγούν σε ναυπήγηση σκαφών. Έχουν προχωρήσει οι πραγματεύσεις. Ναι. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια συνένεση που δεν το έχουμε καταφέρει όμως. Ακόμα, όμως η αρχική πρόταση ήταν η απαγόρευση των επιδοτήσεων που σας ανέφερα ε, για την κατασκευή σκαφών, όχι την δημιουργία νέας ικανότητας. Και τώρα βλέπετε προτάσεις για επιδοτήσεις ε, για την αυπήγηση πλοίων 40 ε, μέτρων. Εγώ δεν βλέπω πως αυτό συνάδει με το στόχο μας. Και επειδή το ανέφερε ο κύριος ε, Μιγιάν Μον, και εμείς θέλουμε και γνωρίζουμε μάλλον πολύ καλά ότι πρέπει να λάβουμε πλήρως υπόψη και τις ανάγκες των αλλιέων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Συμφωνώ απολύτω. Αν θέλουμε να προσελκύσουμε και τη νέα γενιά, δεν είναι διατεθειμένοι να εργαστούν υπό τι συνθήκες που εργάζονταν οι γονεί τους. Και στην περιοχή την οποία κατάγομαι έχουμε πολλά μικρά αλευτικά σκάφη. Ξέρω ποιε είναι οι συνθήκες. Αλλά λέω, μπορούμε να βελτιώσουμε ε, τις συνθήκες, μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, την ασφάλεια, χωρίς όμως να δώσουμε χρήματα για την ε, ναυπήγηση νοσκαφών. Αυτό ήθελα να πω. Κυρία Κόντε. Ε, κύριε Διευθύντα, ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ και που μας δίνετε τη δυνατότητα του διαλόγου, ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες ε, αλλαγές ε, σε θέματα διαχείρισης. Ε, τρία θέματα μας έχουν κληροδοτηθεί από την προηγούμενη θητεία, από το προηγούμενο κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ανησυχίες. Αναφέρομαι κυρίως στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρίως για μικρά ψάρια στην Αντριατική. Ε, μερικοί έχουν μιλήσει για ένα πιάνο ζόμπι, ένα σχέδιο ζόμπι. Οι συνάδελφοι που δούλεψαν πριν από μένα για το θέμα αυτό ε, δεν λένε ότι δεν υπάρχει καμία συνέχεια, δεν εξηγείται η γραμμή που θέλετε να ακολουθήσετε. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω πώς ακριβώς προτίθεστε να προχωρήσετε. Και μία, κάτι άλλο, αυτό ήταν μια ερώτηση, κάτι άλλο. Αναφερθήκατε σε κλιματικές αλλαγές. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω κατά πόσον η Κομισιόν προτίθεται να εκταμιεύσει κονδύλια για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, κυρίως για τα μικρά ψάρια λαμβάνοντας ε, κυρίως υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και οικονομική βιωσιμότητα. Και όσον αφορά τον κανονισμό για τον έλεγχο, θα ήθελα να πω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να προβλέπεται ικανοποιητική οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο, κυρίως για να στηριχτούν οι μικροί αλείς. Και θέλω λοιπόν να πω το εξή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε με απόλυτη σαφήνεια και με απόλυτη πλειοψηφία. Το Συμβούλιο φαίνεται ότι δεν που στασιοποιείται από αυτά που είχαν ψηφιστεί στην προηγούμενη περίοδο. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία μείωση του 4,6% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο ταμείο. Ίσως λοιπόν δεν θα ήταν λάθος, τουλάχιστον λάθος, να ε, προταθεί μία πρόταση διαφορετική από αυτή που είχε ψηφιστεί στην προηγούμενη θητεία. Αυτά ήθελα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Για την Αδριατική, η τροπή που έλαβαν οι συζητήσει τελικά ήταν πολύ ενισχυτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή δεν σεβόταν αυτή η συζήτηση την κοινή ελευτική πολιτική. Οδηγούσε σε μία συνέχιση της επηραλίευσης. Δεν είχε να κάνει με το γάβρο, γιατί σε αυτή την περίπτωση τα μικρά πελαγικά είδη ήταν ο γάβρος και η σαρδέλα, αλλά η συζήτηση που είχε γίνει στην προηγούμενη επιτροπή ήταν η ανάμεξη των δύο. Και αυτό θα συνέχιζε την υπεραλίευση. Κανένας από τους βασικούς κανόνες ε, της κοινή ελευθερικής πολιτικής δεν ε, μπορούσε να τηρηθεί με αυτόν τον τρόπο. Τελικά οδηγηθήκαμε στην Επιτροπή για τη Μεσόγειο, το GFCM. Εκεί συμφωνήθηκαν κατά κατεπήγοντα μέτρα και πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε με τέτοιου είδους μέτρα και στα επόμενα χρόνια. Και το πολιετές σχέδιο για την Αδριατική μπορεί να επανέλθουμε όταν είναι καλύτερες συνθήκες. Όμως, η κατεύθυνση ήταν πολύ ενισχυτική και αντίθετη με αυτό που θέλαμε. Κλιματική αλλαγή τώρα. Όπως είπα στο ΕΤΘΑ έχουμε πει ότι λέω 30% των πόρων θα διοχετευθεί προς δραστηριότητε που θα μετριάσουν την κλιματική αλλαγή. Αυτό ήταν 25% στην πρώτη ανάγνωση, στη θέση μας στην πρώτη ανάγνωση. Μετά, κανονισμούς περιελέγχων. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, αλλά σήμερα ακόμα και, η αεριστεχνική αλληλεία, η μικρής κλίμακας αλληλεία, τα σκάφη κάτω των 12 μέτρων δηλαδή, που δεν ε, χρησιμοποιούν συγκεκριμένο εξοπλισμό. Και πάλι μπορούμε να ελέγξουμε με κινητές συσκευές τα αλλιεύματα. Με άλλους τρόπους λοιπόν που δεν αποτελούν ε, φόρτο. Όμως πρέπει και οι μικρές κλίμακας να αναφέρουν τι αλλιεύουν και πού. Και να αναφέρουν λοιπόν τις δραστηριότητε στη θάλασσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλύπτεται το 100% για την ε, διαμόρφωση αυτής της δυνατότητας καταγραφής. Λοιπόν, οι μικρή κλίμακα ε, αλία σήμερα έχουν ε, εξαιρέσει. Δεν χρειάζεται να καταγράφουν τα λεύματά ναι. τους. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακριβή τους θέση. Μετά, ας δούμε τη Μεσόγειο. Πάνω από το 80% του στόλου στη Μεσόγειο είναι μικρής κλίμακας. Παράκτια αλία Συνήθως λέμε ότι το μικρές κλίμακε είναι και το καλό, το πιο βιώσιμο. Αλλά δείτε την κατάσταση των αποθεμάτων. Υπάρχει τρομερή υπεραλίευση. Εν μέρη επειδή έχουν λάβει εξαίρεση για τα πάντα. Δεν χρειάζεται να καταγράφουν τα αλλιεύματά τους. Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ούτε οι επιστήμονες γνωρίζουν. Κάτι πρέπει να αλλάξει λοιπόν. Ναι, δεν θέλουμε να τους επιβάλλουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις ίδιες που έχουν οι μεγάλοι του κλάδου. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταγράψει κανείς ε, τα λεύματά του, ακόμα και αν έχει ένα μικρό σκάφος. Αλλιώς φτάνουμε σε αυτά που βλέπουμε στη Μεσόγειο σήμερα, υπεραλίευση παντού. Και εγώ δεν μιλάω για το Μαρόκο και τους άλλους, μιλάω για τα ενωσιακά ύδατα τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να το φορτώσουμε σε άλλους. Αυτό θέλουμε εμείς να κάνουμε. Και πάλι θα υπάρχει 100% χρηματοδότηση για τα ε, σκάφη μικρή κλίμακα. Εντάξει, καλύπτουμε πολλά θέματα, αλλά χάνουμε, ε, πάλι περνά και ο χρόνο. Κυρία Τόματσιτ. Eh, eh, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μασάδο για την παρουσία του εδώ. Νομίζω ότι έχουμε σαφείς επιστημονικές ενδείξεις ότι το απόθεμα έχει αυξηθεί ε, περισσότερο, όχι τόσο, περισσότερο στις αρδέλες. παρά στην Ατζούγια πιο συγκεκριμένα. Αυτό δεν ξέρω αν η ΓΑΜΑ δηλαδή εξακολουθεί να προτείνει την εισαγωγή ποσόστοση για τα μικρά πελαγικά στην Αδριατική ή έχουμε κάποια εναλλακτική ε, προσέγγιση. Επίσης, ε, για τα πολιετή σχέδια διαχείρισης, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουμε για τις νέες προτάσεις πολιετών, ε, ιδιαίτερα προφανώς αναφέρομαι στην Αδριατική. Και επίσης ποια είναι τα οι προθέσει μας ε, για τα πολιετή, για τα υπόλοιπα είδη στην Αδριατική. Ο κύριο Περέιρα, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ το Γενικό Διευθυντή. Ε, αναφερθήκατε στις θετικές εξελίξεις ε, σχετικά με μια σειρά από είδη. μιλήσατε και για αριθμούς ρεκόρ τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμπεράνει έτσι ε, ότι η, κατάσταση είναι θετική συνολικά στον κλάδο, συνολικά στο πεδίο. Ιδιαίτερα στην βιοτεχνική και μικρή κλίμακα η αλληλεία η κατάσταση είναι οτιδήποτε εκτός από ε, θετική και ευίωνη. Πρόκειται για μια βαθύτατη κρίση Επίσης ε, μα είπατε ότι πρέπει να σκεφτούμε ε, πέραν της αλληλείας. Ε, δίκαιο έχετε, αλλά η πολιτική αλληλείας είναι μια από τις παλαιότερες και από τις λίγες κοινέ πολιτικές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα. Μπορεί κανείς να προσπαθήσει να ξεπεράσει και την εντολή του, αλλά προς, τουλάχιστον πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τα ελάχιστα στον προπολογισμό για να εκτελέσουμε, να υλοποιήσουμε την ίδια την πολιτική. Δεν έχουμε μία, ενώ έχουμε στην ουσία μία ε, κάπη η οποία υποχρηματοδοτείται. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον άλλων περιοχών, αλλά χρειαζόμαστε τους πόρους που χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε την κοινή αλληλευτική πολιτική γιατί η αλληλεία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποκλειστική, δεν μιλούμε καν για μεικτή. Και έχουμε συστηματική υποχρηματοδοτήση τη πολιτική και του τομέα, το οποίο μου οδηγεί στο EMFF. Εδώ κύριε Γενική Διευθυντά, η Κομισιόν πρέπει να είναι πιο ανοιχτή. Είναι το μόνο που μπορώ να σα πω. Ε, πιο ευέλικτη. Λιγότερο έτσι ε, πα, ε, αποκρισταλωμένη, παγιωμένη και περιχαρακωμένη στις θέσεις τη τα όσα ε, υιοθέτησε το, το Κοινοβουλίο δεν μας οδηγούν στο πέρασμα της ε, δυνατότητα. δυνατότητας. Δεν πρέπει να φοβίζουμε τα νέα μέλη λέγοντας τέτοια πράγματα. Αυτή η, θέση ε, ε, ενεκρίθη με πολύ μεγάλη πλειοψηφία διαφόρων πολιτικών ομάδων και δεν θα οδηγήσει σε υπερβολική ε, δυνατότητα. Εάν η Κομισιόν έχει πράγματι αυτή την ανησυχία, πράγματι, τεχνικά και επιστημονικά, θα πρέπει να προτείνει πράγματα ε, προσαρμογής, αν θέλετε, του πλαισίου στο οποίο έχει τοποθετηθεί και το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν δεν θέλει να αποτρέψει επενδύσεις για την καλύτερη ασφάλεια ε, και την καλύτερη ε, ζωή των αλλιέων επί των σκαφών έχουμε μιλήσει για την, την κατάσταση παλαιών σκαφών τα οποία δεν μπορούν να βελτιωθούν έτσι όπως εσείς προτείνετε. Και το, και το τελευταίο σημείο, Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξή. Μπορείτε να μας δώσετε μία επικαιροποίηση για τις ε, παραβάσεις ε, και για την αναστολή πληρωμών ε, ως αποτέλεσμα ελέγχων υπάρχει κάτι τέτοιο που να συμβαίνει ή όλα αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Και τελευταίο ερώτημα για τις ε, σαρδέλες. Όχι, όχι λέει ο πρόεδρος σας παρακαλώ. πολύ πρόσφατα είχα εκδηλώσει την ανησυχία μου αυτού, δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη αυτό για την αύξηση στην βιομάζα, στο απόθεμα, στην συγκεκριμένη περιοχή. Πολλά ερωτήματα λέει ο πρόεδρος, τα οποία τα βάλαμε έτσι, τα υπερσυμπιέσαμε σε πολύ μικρό χρόνο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό κύριε Πρέ. Μήπως ε, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε πρώτα όλα τα ερωτήματα και μετά να δοθεί συνολικά μία απάντηση. Γιατί περνάει η ώρα και δεν έχουμε χρόνο να θέσουμε όλα τα ερωτήματά μας, δεν έχουμε και συχνά την ευκαιρία να τα θέσουμε. Ναι, αλλά εσείς θα πάρετε το λόγο μετά, ακριβώς μετά. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στο Γενικό Διευθυντή. Thank you. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, οι επιστήμονες μας λένε ότι ο όγκος έχει αυξηθεί στην Αδριατική. Είναι κάτι που πρέπει να δούμε πολύ πολύ προσεκτικά. Ε, ε, εμάς η μόνη μας πρόθεση είναι να εργαστούμε εντός του πλαισίου του GFC. Και η κυρία Τόματσικ το ξέρετε και το έχουμε πει και στο παρελθόν. Ε, στη Μεσόγειο δεν μπορούμε να έχουμε τάκο που έχουμε σε άλλες θάλασσες. Αλλά και στην Ατζούγια και στη Σαρδέλα είχαμε πρόβλημα στη Βυσκαϊκή γιατί εισήχθησαν τάκ και το απόθεμα αποκαταστάθηκε. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Μεσόγειος είναι τόσο διαφορετική και δεν μπορείτε εκεί να έχετε τάκ. Προς το παρόν εργαζόμαστε στο πλαίσιο του GFCM και εξετάζουμε εσωτερικά τι μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει απόφαση. Υπάρχουν ε, περιφέρειες, ζώνες και είδη που θα πρέπει να καλυφθούν από πολιετή σχέδια. Έχετε δίκιο. Τώρα κύριε Φερέρα γνωρίζω ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια στους διάφορους υποκλάδους αλλά είχαμε μια συνολική κερδοφορία με ε, τις τάξεις του 80%. 18-19% ε, με συγχωρείτε. Το οποίο δεν είναι άσχημο. Γνωρίζετε πώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν. Και στο IMF e υπάρχει χρηματοδότηση για την κλιματική αλλαγή, για του μπλε στόχου. αλλά ε, ε, εντάσσονται στους στόχους ε, τη της διαχείρισης. Άμεσης δηλαδή διαχείριση. Και αυτό το χειρίζεται η Κομισιόν. Αν θέλετε να πάτε σε αυτή την περιοχή, που εγώ πιστεύω ότι πράγματι θα πρέπει να πάμε, τότε θα πρέπει να έχουμε τους φακέλους άμεσης διαχείρισης να τους αυξήσουμε ελαφρά. Και οι, οι πόροι, τα αποθέματα των ειδών μετακινούνται αλλού με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να έχουμε ευρύτερη εικόνα δηλαδή. Γιατί αποφασίζει κανείς τάκ, πάει μετά στη θάλασσα και έχουν φύγει τα ψάρια. Ναι, έχετε δίκιο ότι η Κομισιόν πρέπει να είναι πιο. να μην είναι τόσο άκαμπτη. Ενδεχομένω, αλλά. Θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση αυξημένη δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δούμε στου μερίδια διαλόγου πώ μπορούμε να αντισταθμίσουμε αυτό το κίνδυνο. Για τη Σαρδέλα. Τέλο. Είχα πει και σε μια συνέντευξη ότι το απόθεμα βρίσκεται σε κατάσταση κακή. Εγώ δεν είπα εκεί ότι πρέπει να έχουμε κι άλλη μείωση. Είπα ότι το απόθεμα είναι ευαίσθητο. Τώρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ε, ισχυρίζονται διάφορα πράγματα για συγκεκριμένες περιοχές ε, σαρδέλας. Ας τα δούμε στην ISIS και επανερχόμαστε. Λοιπόν, όσον αφορά τη διαχείριση χρόνου, δεν νομίζω ότι τα πάω και πάρα πολύ καλά. Τώρα, ε, τα μέλη. Για ένα λεπτό παρακαλώ να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Να έχω ένα ερώτημα από τις κάτω χώρες ό,τι αφορά την ε, υποχρέωση εκφόρτωσης και τις εξαιρέσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση ε, στις εξαιρέσεις Σε ό,τι αφορά λοιπόν την υποχρέωση εκφόρτωση, ε, τα πράγματα είναι ιδιαίτερα στι 10 χώρε. Δεν έχει καμία ιδέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι η πρακτική. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό σύστημα στην ε, χώρα μου, αλλά φαίνεται ότι απαγορεύεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή. Δεν γίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Πρέπει να πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει πώ λειτουργεί το Ολλανδικό σύστημα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στη ζήγηση των ε, ψαριών που φτάνουν για ε, κατανάλωση, αλλά παράλληλα υπάρχει και το σύστημα με τον ε, πάγο, αλλά και πάλι υπάρχει ποικιλία ε, της ποιότητας, διαφορές στην ποιότητα του πάγου. Αν όμως ένας έμπορος δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Ναι, το ερώτημα λοιπόν. Αυτό δεν ισχύει για την Ολλανδία, για όλη την Ευρώπη. Ένα παράδειγμα μου. Εγώ είμαι και πλήρες μέλο, έτσι, γιατί άλλοι μίλησαν πριν που δεν ήταν. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, τα σημεία πώληση σε όλη την Ευρώπη, θα ήθελα να τα εξετάσετε όχι μόνο για τις κάτω να αρχίσουμε λοιπόν να δούμε και τις εξαιρεσει. Mr. Ευχαριστώ. Σύντομα δύο παρατηρήσεις. Ε, μιλήσατε για την ε, παραγωγή ενέργεια στη θάλασσα. το αναφέρατε ως ε, ευκαιρία. Από ό,τι βλέπω όμω υπάρχει και σημαντική απειλή για την αλία. Αν δείτε τη Βόρεια Θάλασσα, για παράδειγμα. Έχουμε περίπου 22.000 ε, αναμογεννήτριε. Το 1 τέταρτο λοιπόν τη Βόρεια Θάλασσα είναι γεμάτο με αναμογεννήτριε. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εθνική ε, αναγκαιότητα, αυτό είναι γνωστό, αλλά από εκεί και πέρα, πόσο, εμπλέκονται εδώ, πόσο εμπλέκεται εδώ η DG Mare, μήπως θα πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα για το τι σημαίνει αυτό για την αλληλεία. Αυτά τα μεγαλεπίβολα σχέδια, τι θα σημάνουν για την αλληλεία. Για να έχουμε πιο ρεαλιστικές προσδοκίες. δεύτερον, υποχρέωση εκφόρτωσης. Ε, μας ε, φτάνουν πολλές καταγγελίες για το σύστημα σίγουρα υπάρχει ένα πλαίσιο σχέση με τα τεχνικά μέτρα, αλλά ε, πρέπει να υπάρχει πραγματικά μία αξιολόγηση ε, και μάλιστα σύντομα. Πότε προβλέπετε να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Mr. D'Amato. <coughs> Mr. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ερωτήσεις. Ε, από τη μια δεν έχουμε μελέτες που να αφορούν ε, στη μείωση των αποθεμάτων. Έχουμε όμως μελέτες ε, για τις ζημιές που προκύπτουν από τη ρήπανση. Έχουμε στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει υπερβολική ε, μετακίνηση των σκαφών ή επίσης και για τους αγωγούς. Τα κατά την άποψή μα, είναι τα βασικότερα αίτια και αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τώρα, όσον αφορά την υποχρέωση εκφόρτηση, νομίζω ότι δουλέψαμε για το ΦΕΠ στην προηγούμενη θητεία και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμφωνήσει ότι πρέπει να υπάρχει ειδική ενίσχυση για τα μικρά ψάρια και κυρίως για την διατήρηση και επιβίωση των αλλιέων. Θέλω να ρωτήσω. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και τέλος, ε, θα ήθελα να υποβάλω μία πρόταση. Ε, έχοντας κατά νου ε, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία, θα θυμάστε ότι όσον αφορά τα οποροκυπευτικά και το γάλα, υπήρχε ένα πρόγραμμα να χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Γιατί να μην υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που να αφορά στα ψάρια, να γίνει και με τα ψάρια, ακριβώς το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις τελευταίες εκλογές ε, το κόμμα υπέρ του Brexit κέρδισε την πλειοψηφία, ο κύριος ε, Γενικός Διευθυντής θα δεχτεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το δικαίωμα να είναι ανεξάρτητο κράτος, ε, παράκτιο κράτος και μετά το Brexit. Επίσης, ο κύριος Διευθυντής θα αναγνωρίσει ότι η Βρετανική αλληλεία πρέπει να είναι εξάρτητη, κανείς δεν να παρεμβαίνει και μόνο η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει το δικαίωμα να αναδιανύμει τις ε, δυνατότητες αλληλείας ε, στα δικά της ε, τα ίδια, ενώ παλαιότερα αυτό ίσχυε για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για να τα καταλάβετε καλύτερα, έχω ένα φυλάδιο για σας κύριε Διευθυντά, για σας κύριε Πρόεδρε και είχα και ένα και για τον κύριο Βαντάλεν για να τα καταλάβετε όλα καλύτερα. Θα σας δώσω αυτά τα φυλάδια στο τέλος. Ευχαριστώ τον κύριο Γενικό Διευθυντή για την παρουσία του και πολύ χαίρομαι που στην παρέμβασή σας ε, αναφερθήκατε στις προκλήσεις όχι μόνο για την αλληλεία αλλά συνολικά για τους ωκεανούς, για τη γνώση, για την συντήρηση, για την προστασία των πορών της μπλε οικονομίας, της διακυβέρνησης. Εγώ είμαι νέο μέλος του Κοινοβουλίου και συμμύριζομαι μαζί σας ε, τον ρόλο που μπορεί να διαματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο των θαλασσών και της αλλιευτικής δραστηριότητας αναφερθήκατε και στο Green Deal μεταξύ άλλων και της φιλοδοξίας που πρέπει να έχει η Κομισιόν και η ερώτηση μου είναι τελικώς πώς μπορεί η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές ναι, για να γίνει και γεωστρατηγικά αν θέλετε παίκτη στα θέματα της αλληλείας και της προστασίας του περιβάλλοντος ε, να, να έχει τη θέση που της αναλογεί αν θέλετε σε παγκόσμια κλίμακα. Ευχαριστώ ο κύριος Γενικός Διευθυντής παρακαλώ να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για την κυρία Σχάιερ για τις υποχρεώσεις ε, εκφόρτωσης. Ε, είναι σημαντική πρόκληση, πρόβλημα για τον κλάδο και για τις αρχές ως προς τον έλεγχο. Οι εξαιρέσεις που παρέχονται, και πάλι λέω, ε, οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν με συναπόφαση και με τους συνομοθέτες, αλλά με την απόφαση την τελευταία έγινε ακόμη πιο δύσκολο να ελέγξουμε. Καταρχάς, για τον δίκτυ επιβίωσης του ε, αποθέματος. Όταν φορτώνεται και όταν απορρίπτεται. Για το ελάχιστο μέγεθος. Που δεν πρέπει κανείς να αλλιεύει, δηλαδή πολύ μικρά ψάρια. Αν θέλει κανείς να έχει μόνο 5% κάτω του ορίου, ε, όταν εισέρχεσαι στο λιμένα. Αλλά στην πράξη, πώς επιλογίζει κανείς το 5% στη θάλασσα από όλα αυτά που αλλιεύει. Πώς γίνεται αυτό στην πράξη, πώς το κάνεις. Πρόκειται για ένα πρόβλημα τεράστιο. Ε, έρχονται στους λιμένες τα σκάφη και δεν ξέρει κανείς αν έχουν απορρίψει στη θάλασσα ή τι έχουν κάνει. Και η ενδείξει που έχουμε εμεί στη διάθεσή μα είναι ότι η απόρριψη συνεχίζεται. Χωρί έλεγχο, πώ να ξέρετε τι έχει υλοποιηθεί. Τι διατάξει όμω τι έχει ο βασικό κανονισμό. Και μπορούν επομένω να τι χρησιμοποιήσουν οι αλλοί. Ε, ένα από τα σημεία βασικότερης ανησυχίας είναι η καλύτερη οργάνωση του θαλασσίου χώρου. Γιατί αναφερθήκατε σαν αιμογεννήτριες. Είναι αλήθεια ότι θα έχουμε μεγαλύτερη δραστηριότητα στη θάλασσα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να την οργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Χωροτακτικά δηλαδή, ε, ούτω ή πρέπει να οργανώσουμε το θαλάσσιο χώρο. Γιατί αυτά θα γίνουν. Και βεβαίως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις ε, ε, πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα και τα λοιπά. Και την εξόριξη σε, σε βαθία ύδατα. Ε, μην ξεχνούμε ότι για πρώτη φορά, για πρώτη φορά στο νέο Horizon θα έχουμε τη μία από τις αποστολές με ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τους ωκεανούς. Την οποία θα ηγείται ο Πασκάλα Μη. Δηλαδή υπό το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρώπης έχουμε μία από τις αποστολές που αναφέρει του ωκεανούς. Και οπωσδήποτε θα, εκεί θα προσπαθήσουμε να αναφερθούμε στα προβλήματα που και εσείς αναφερθήκατε, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα είναι παράκτιο κράτος <laughs> όταν αποχωρήσει όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε όταν ανοίξουν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο προς το παρόν. Ελπίζομαι απλώς ότι θα μπορέσει να εξέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο με τρόπο μη άτακτο. Και, και κυρία Σαπό, η, η Ηνωμένη Ευρώπη το γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε, είναι ήδη μια μεγάλη αλλιευτική δύναμη αλλά πρέπει να προσέχουμε να διαχειριζόμαστε το πεδίο αυτό όσο καλύτερα μπορούμε. Αν θέλουμε να ταΐσουμε τον, τον πληθυσμό που εκτιμάται πλέον στα 9 δισεκατομμύρια, γνωρίζετε τις παραγωγές διοξιδίου του άνθρακα που υπάρχουν, η εναλλακτική ελιευτική έχει εναλλακτικέ ε, δυνατότητες αλλά ε, ούτε θέλουμε και ούτε μπορούμε να έχουμε ε, χώρους υδατοκαλλιέργεια οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Προσοχή. Μέτρο και καλή οργάνωση. Αν δούμε την ζημιά που έχουμε κάνει συνολικά στον πλανήτη, την ορατή ζημιά, χερσαία τουλάχιστον, που δεν μας απέτρεψε ε, να προβούμε σε μεγάλες καταστροφές φυσικές, στον ωκεανό δεν το βλέπουμε. Δεν φαίνεται η ζημιά τόσο εύκολα. Αλλά είναι τεράστια η ζημιά και πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί με το θαλάσσιο περιβάλλον. Ε, κυρία Ταντία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Εσείς είπατε ότι το 80% των αποθεμάτων στη Μεσόγειο είναι πλεόνασμα ε, και το είπατε και το επαναλάβατε στις απαντήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν τα στοιχεία αυτά ε, μπορούμε ή μάλλον το πω αλλιώ, πού αναφέρονται ακριβώς αυτά τα στοιχεία, γιατί αναφέρθηκε επίση ότι τουλάχιστον στη Μεσόγειο ε, δίδονται συγκεκριμένες, περιορισμένες άδειε. Οι ε, ψαράδες, οι ελίες μα λένε κάτι τελείω διαφορετικό, ότι δεν υπάρχουν, υπάρχει ε, έλλειψη ψαριών στη Μεσόγειο. Και όσον αφορά την ερώτηση από τη Σνάλφο Φερέιρα, μιλήσατε για μικρό τζίρο. Μήπως μπορείτε να μας πείτε σε ποιες ε, περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεστε. Γιατί στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, ε, καταραίει νομίζω η Ελία και το ίδιο περίπου ισχύει και για την Πορτογαλία. Ε, παρακαλώ, εσείς πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά που είπατε και θα ήθελα να πω ότι στην απάντησή σας είπατε δεν θέλετε να ε, τρομάξετε ένα μέλη. Εγώ είμαι νέο και δεν τρόμαξα. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Αναφερθήκατε στις ε, στην εφαρμογή σε ένα σύγχρονο τρόπο ε, εφαρμογής. Μιλάτε για το CCTV και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι οι Σκοτσέζοι αλληλείς είχαν αυτά τα κλειστά κυκλώματα, το CCTV, εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό δεν είναι σύγχρονο, ούτε κάτι καινούριο. Άλλο κατάλογο ε, καινοτομιών να μας παρουσιάσετε. Το δεύτερο, για το Brexit. Λυπάμαι. Κοιτάξτε, έχει τελειώσει η ώρα. Δεν θα, απλά δεν θα σας απαντήσει ο διευθυντής. Παρακαλώ. μετά πάμε έξω από την αίθουσα αν θέλετε να τα πούμε. Να σας πω λοιπόν ότι η πρόθεσή μου δεν ήταν να πω ότι <laughs> το κλειστό κύκλωμα θα είναι η ναυαρχίδα των ε, καινοτομιών. Υπάρχουν και άλλα πράγματα ε, που είναι καινοτόμα, όπως ε, ας πούμε τα κινητά τηλέφωνα. Ε, τώρα όλα γίνονται με χαρτί και όλα αυτά είναι πολύ βαριά. Υπάρχουν λοιπόν καινοτομίε που δεν θα είναι μόνο κλειστά κυκλώματα και έτσι να μπορεί κανείς να κάνει πραγματική καταγραφή των αλληλευμάτων. Σε αυτό βασικά αναφερόμουν. Αλλά σε διμερές επίπεδο μπορούμε μετά να συζητήσουμε. Λοιπόν, στην δική σας την ερώτηση, κυρία Ταντίν, ε, εγώ δεν λέω ότι ε, το 86% αναφέρεται ένα στοιχείο για την αλληλεία για το 86%. Εγώ δεν το είπα εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Αν θέλετε μετά ε, μπορούμε να το ξαναδούμε. 15 χρόνια ε, εδώ πάντα επέκρινα τους προέδρους που δεν έκαναν καλή διαχείριση χρόνου. Να και εγώ που το ίδιο μου συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, ε, καλύψαμε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθύντα. Πότε φεύγετε? Τον Οκτώβριο. Ελπίζω να μην πάρετε και την αδειά σας ε, και να μπορέσετε μέχρι τότε να εργαστείτε. Τα ξαναλέμε στις 2.30.